So, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Zu unterhalten oder, oder hier ruhig Ihre Plätze einzunehmen. Καθίστε παρακαλώ ή αν θέλετε να συνεχίσετε τα πηγαδάκια σας παρακαλώ να περάσετε έξω. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες ε, τώρα, πάνελ 1. Όπως ξέρετε, το πάνελ αυτό ε, έχει προσκληθεί για να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην έκθεση που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες εδώ τους οποίους είχαμε επιλέξει και σήμερα είναι εδώ παρέντες. Καταρχάς, Πρόεδρος αναρωτιέται μήπως δεν δουλεύει η διερμηνία, αλλά όλα δουλεύουν καλά. Έλεγα λοιπόν Έχουμε έξι μέλη στην Επιτροπή Εμπειρονοχωνομόνων, δυστυχώς έχουμε μόνο τους τρει εδώ σήμερα, αλλά και οι έξι μας έχουν δώσει γραπτή έκθεση επί του θέματος. Και έχουμε ένα έγγραφο το οποίο ετοίμασε το τμήμα πολιτικής Α. Στην πρώτη έκθεση ο καθηγητής Κάμπος Εκούνια, καθηγητής ε, του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, Πανεπιστημίου Νόβα της Λισαβόνας έχει φέρει ένα τμήμα της εκθεσής του, το οποίο θα διανύμουμε σε όλους. Έχουμε λοιπόν, όπως σας έλεγα, τρεις προσκεκλημένους εδώ, τον καθηγητή Κάμπος Εκούνια, καθηγητή της της Νόβα της Λισαβόνας, κατόπιν τον Λορέντσο Ντεάντζελης, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βενετίας και τέλος τον κύριο Σόνι Καπόρ. διευθύνοντα σύμβολα μια επιχείρησης η οποία είναι γνωστή με το όνομα Redefine και τον έχουμε ξαναδεί εδώ. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Κάμπο Σεκούνια. Θα ήθελα να σας ζητήσω να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την παρέμβασή σας και να εστιάσετε σε 10 λεπτά ή και λιγότερο στα θέματα που σας απασχολούν. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd uh, like to say that it... Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ. Πολλές φορές συμμετείχα στα ΕΚΟΦΗΝ, στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Έχω έρθει στις Βρυξέλλες και στα θεσμικά όργανα πολλές φορές, αλλά πρώτη φορά βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μεγάλη μου χαρά και είναι πρώτη φορά που βλέπω τις Βρυξέλλες με ήλιο μία ηλιόλουστη μέρα, σπάνιο φαινόμενο. Έχω ορισμένα σχόλια γενικής εμβέλειας, τα οποία θα διανεμηθούν σε ένα λεπτό και άλλα στοιχεία που θα βάλω στην τελική έκθεση. Το έγγραφο θίγει αρκετά ζητήματα για την αντιμετώπιση των θεμάτων, είναι προκλητικό και μιλά για την μεγάλη αυτή ύφεση που διανύουμε. Και σκόπιμο είναι να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε μία άλλη μελλοντική κρίση, ενδεχόμενη κρίση. Θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι το έγγραφο θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή ε, σε μία ανάλυση των αιτίων της μεγάλης ύφεσης να ε, δει δηλαδή τα αίτια του κακού καθώς και, τα, και μια πολιτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης, η πολιτική αυτή θα πρέπει να αφορά μια σαφή στοχοθέτηση, κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντα και πολλές φορές έχουμε συστάσεις ε, ευρείας εμβέλειας που έχουν, στόχο, ε, που έχουν έναν πολλαπλό στόχο θα μπορούσα να πω. Σε αυτή την περίπτωση τα αίτια σχετίζονται και με ορισμένες παρενέργειες θα μπορούσα να πω ως προς τη μεγάλη αυτή ύφεση, δηλαδή την κατανομή του εισοδήματος, θέματα περιβαλλοντικά και τα δύο αυτά ζητήματα θα πρέπει να φορούν ξεχωριστές συνεκτικές πολιτικές και να μην ε, προσμιγνύονται με ε, την, ε, το ειδικό ζήτημα της μεγάλης αυτής ύφεσης. Δηλαδή να μην υπάρχει σύγχυση στόχων και πολιτικών. Δεν είναι και πολύ καλή ιδέα εκ προημίου. Νομίζω ότι το έγγραφο παρουσιάζει μια προσέγγιση που είναι αρκετά επικεντρωμένη και δεν αφήνει χώρο για εθνικές πολιτικές. Επίσης προσπαθεί να ε, ε, ξέβρει μία ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Υπάρχει μία ανισότητα, μία ανισορροπία η οποία όμως ε, δεν είναι βιώσιμη θα πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδιαίτερα ως προς τις ε, φορολογικές πολιτικές, οι οποίες δεν πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο αποκλειστικά. Επίσης, το έγγραφο στυλιτεύει και θέτει ευθύνες, δηλαδή ε, μιλά για τις αγορές, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ έχω διαφορετική προσέγγιση. Δεν κατακρίνω μόνο τις αγορές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιρρύψουμε την ευθύνη στις εθνικές κυβερνήσεις περισσότερο. Επίσης, το έγγραφο αναφέρει την ενδεχόμενη εναρμόνιση πολιτικών σε ορισμένους φορείς συμφωνώ ως προς την φορολογική πολιτική, η οποία πρέπει να είναι πιο εναρμονισμένη, ε, ιδιαίτερα ως προς την ε, φορολόγηση του κεφαλαίου. Δεν ξέρω ως προς τα ελάχιστα ημερομίσθια ή τους ελάχιστους μισθούς, διότι εξαρτώνται από την παραγωγικότητα και μπορεί να σημαίνει αύξηση της ανεργίας, ειδικά στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Άρα η εναρμόνιση πολιτικών θα πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά. Επίσης, ε, ε, γίνεται λόγος για μια πολιτική παρεμβατισμού. Ιδιαίτερα όταν αποτυγχάνει η αγορά και οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, τίνουν προς αυτό. Δηλαδή χρειάζεται μια ρύθμιση αυτών των αγορών αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ρύθμισης, δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις. Εάν δούμε τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι του υπηρετικού συστήματος βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα υπηρετικά ευρωπαϊκά ρυθμιστικά συστήματα είναι πολύ πιο αποδοτικά από το αγγλοσαξονικό σύστημα. Επίσης, ο κρατικός παρεμβατισμός επαφίεται στο κράτος βέβαια, δηλαδή να γίνει μια μελέτη κόστους ωφέλειας ε, χωρίς να γίνει μια ισοπαίδωση των ε, θεμάτων όλων. Ως προς την κατανομή του εισοδήματος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα και κατά την τελευταία δεκαετία, τα 15 τελευταία χρόνια, ε, διευρύνεται αυτό το χάσμα στην Ευρώπη. Δεν ε, ξέρω κατά πόσο το σφάλμα επαφείται στην ε, κρίση. Δεν ξέρω δηλαδή εάν η ύφεση είναι υπέτεια για την ε, κατανομή εισοδήματος. Ίσως η κατανομή εισοδήματος θα πρέπει να είναι ένα θέμα καθο... αυτό καθεαυτό, διότι είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Η ασυμμετρία κατανομής εισοδήματος έχει σχέση με την εξέλιξη της Ινδίας και της Κίνας, που είναι μεγάλοι παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας, γιατί εν μία νυχτή στην ουσία διπλασιάστηκε ο πληθυσμός και έτσι συμπιέστηκαν τα εισοδήματα. Και σε επίπεδο είπα έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα ημερομίσθια. Επίσης υπήρχε άμεση ζήτηση κεφαλαίου με την ε, παρεπόμενη επιστροφή του. Άρα ε, υπήρχε αυτός ο παράγοντας του χάσματος της κατανομής εισοδήματος, αλλά το αντίθετο συνέβη στην ε, ε, Κίνα και την Ινδία. Δηλαδή ότι τα, εκεί τα ημερομίσθια και οι μισθοί ανέβηκαν και αυτό είχε επίπτωση στην κατανομή του κεφαλαίου. Στην Ευρώπη θα πρέπει να δούμε το θέμα της επανακατανομής της ενδεχόμενης αυτής επανακατανομής. Αλλά το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα και την Ινδία. Επανερχόμενο στη μεγάλη ύφεση, θα ήθελα να τονίσω ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχαμε μεγάλες απώλειες κεφαλαίου και μεγάλη αύξηση του δίκτυα ανεργίας. Κάτι το οποίο είχε επιπτώσει στην κατανομή εισοδήματος. Δηλαδή, οι βασικοί χαμένοι ήταν αυτοί που κρατούσαν το κεφάλαιο στα χέρια τους και οι άνεργοι. Αυτοί που κατάφεραν να κρατήσουν την εργασία τους είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που ίσχυε δύο χρόνια πριν. Πολλές φορές η κατανομή εισοδήματο είναι ένα μακροχρόνιο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μακρόπνοες πολιτικές. τα, τα σημερινά προβλήματα αφορούν το ύψος του χρέους ή την μείωση των αποταμιεύσεων σε πολλές χώρες. Η συσσόρευση χρέους από χρηματοπιστωτικά, καταναλωτές κλπ. δημιουργεί συστημικούς κινδύνους που δεν γίνονται αντιληπτοί κατά μία περίοδο ανάπτυξης. Άρα το θέμα των ενυπόθηκων δανείων, των subprimes, δεν ήταν το αίτιο, η αιτία, αλλά έδωσε μία όθηση σε αυτή την κρίση. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τις αποταμιεύσεις, το δίκτυ αποταμιεύσεων που μειώθηκε άρδιν σε πολλές χώρες και νομίζω ότι αυτό το έγγραφο ασχολείται με αυτό το θέμα του χρέους ή του δίκτυ αποταμιεύσεων κατά πολύ κατακαιρματισμένο τρόπο, ενώ θα πρέπει να είναι η, εμπροστοφυλακή των πολιτικών μας. Έχω στοιχεία για το 95-91-2007 στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ και στη Γαλλία και τη Γερμανία βλέπουμε ότι τα τελευταία 13 ε, χρόνια ο δείκτης αποταμίευσης ήταν 15 με 16%. Η Πορτογαλία έπεσε από 13% το στο 6% το 2007. Η Ισπανία από 17,5% σε 10% το 2007 και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο από 10% σε 2% το 2007 σε σχέση με το 1995. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα για να αντιμετωπίσουν ε, τη μεγάλη ύφεση είναι οι χώρες όπου έχει πέσει κατά πολύ ο δείκτης αποταμίευσης. Δηλαδή στη Γερμανία βλέπουμε ότι οι χώρες που αντιμετωπίζουν καλύτερα την ύφεση έχουν και υψηλότερο δείκτη αποταμιεύσεων. Και αυτό επεξηγεί και το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην Ισπανία και την Πορτογαλία διότι ο μειούμενος δείκτης αποταμιεύσεων ή ο χαμηλός δείκτης αποταμιεύσεων οδηγεί στα μεγάλα ε, λογιστικά ελλείμματα. Και αυτό σημαίνει για τις αγορές απώλεια ανταγωνιστικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια, με συγχωρείτε, το 2008-2009, τη στιγμή που οι δείκτες αποταμίευσης ε, αυξήθηκαν σε πολλές χώρες, ε, τα καταφέραμε πολύ καλά και με την ανταγωνιστικότητα. Ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ε, βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο του ευρώ. Ένα άλλο ζωτικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στο έγγραφο είναι η διαφάνεια φορολογικών στοιχείων. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε τις αποταμιεύσεις του δημόσιου τομέα. Δεν έχει νόημα να ενισχύσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης εάν δεν είμαστε πιο αποδοτικοί και διαφανή στη φορολογική πολιτική και υπάρχουν πολλοί τρόποι ωρεοποίησης των λογιστικών στοιχείων, τα οποία έγιναν αποδεκτά από τη Eurostat, ενώ δεν θα έπρεπε. Άρα υπό την ευρία έννοια, μάλλον θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύτερο ορισμό του δημοσίου χρέους και πολλά είδη φορολογικών εσόδων θα πρέπει να αποκλειστούν, ε, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Εν πάση περιπτώσει, η διαφάνεια είναι μια λέξη κλειδί για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε, κύριε Κάμπος δεκούνια Ο κύριος Λορέντζο Ντεάντζελης έχει το λόγο από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μιλήσω Ιταλικά, διότι βλέπω ότι είναι πολύ αποδοτικό το σύστημα της διερμηνίας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Κυρίες και κύριοι, στην έκθεση της κυρίας Περβάνς Περές, η οποία μου δόθηκε προς ανάγνωση και σχολιασμό, να πω εδώ ότι πρόκειται για μια πληρέστατη έκταση. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, σημεία τα οποία φαντάζομαι ότι συμμεριζόμαστε όλοι. Κάποια άλλα τα οποία χρήζουν συζήτηση. Εγώ προσωπικώ έχω επιφυλάξει μόνο για τέσσερα θέματα, δεν τα συμμερίζομαι αυτά και αυτό είναι η δημιουργία ενός corporate tax ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν εταιρικό φόρο. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο σόφρον γιατί είναι αρκετά μεγάλο το φορολογικό άχθος. Και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μετά την εισαγωγή του ευρώ έχουν ε, καταβάλει πολύ μεγάλες συνεισφορές ε, για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Όπως επίσης δεν συμφωνώ και με το σημείο της εισαγωγής φορολόγησης ε, στις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ε, αυτή τη στιγμή ο κλάδος είναι αποδυναμωμένος. Δεν χρειάζεται να δέχεται και άλλα χτυπήματα μέσω νέων φορολογικών επιβαρύνσεων. Και άλλωστε η Goldman Sachs μας δείχνει ότι δεν είναι οι τράπεζες αυτές που δεν κάνουν καλές πολιτικές, αλλά ότι πρέπει να απομακρυνθούν συγκεκριμένοι τραπεζίτες και να τους επιβληθούν φυσικά και κυρώσεις ενδεχομένως. Όλοι αυτοί οι φορές, όπως η Γιάς και ο Γιώσκο, έχουν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουν, τον οποίο διαδραματίζουν εδώ και πάρα πολύ καλά και πριν τους περιορίσουμε την αυτονομία τους, καλό θα ήταν να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Κάποια από τα σημεία τα οποία επισήμανα ε, τα άκουσα και σήμερα το πρωί από τον κύριο Μποργέτζιο, ο οποίος μπόρεσε να διαβάσει την έκθεσή μου λίγο νωρίτερα. Διανέμεται η έκθεση και μπορείτε να την ε, λάβετε υπόψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μποργέτζιο που έλαβε υπόψη του κάποιες από τις απόψεις μου να περάσουμε τώρα απευθείας ε, στην έκθεση. Την έχω χωρίσει σε δύο τμήματα, στα ε, μέτρα διακυβέρνησης και τα μέτρα της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Τα μέτρα της διακυβέρνησης. Υπάρχουν κάποια προφανή μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου όμως θα πρέπει να επισημανθούν εκ νέου όπως για παράδειγμα η μείωση του κόστους ε, της δημόσιας διοίκησης. Η μείωση του κόστους της δημόσιας διοίκησης συνεπάγεται και περισσότερα κονδύλια στην τσέπη των φορολογουμένων που μπορούν είτε να τα χρησιμοποιήσουν για να καταναλώσουν, κυρίως οι οικογένειες, ή για να αυξηθούν οι επενδύσεις για τις επιχειρήσεις. η ανάγκη να μειωθεί το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα, προσοχή εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα, ε, και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με κάθε μέσο ε, είναι πλέον, ε, έχει περάσει τη λύθη φαίνεται, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Επίσης πρέπει να αυξηθεί η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και να αυξηθεί και η επιτήρηση και επίσης να μειώσουμε το φαινόμενο ε, της, ε, των δασμών, της μόχλευσης, της ε, στην, στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερος έλεγχος στον μεγάλο κίνδυνο ρευστότητα. Το επισημένο αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίσουμε ε, τους ε, τίτλους, ομόλογα ή οτιδήποτε άλλο εκδίδονται και είναι ε, υψηλού κινδύνου, ε, είτε είναι από τράπεζες είτε από άλλους φορούς και θα πρέπει οι τίτλοι αυτοί να εκδίδονται από τη δυνατότητα που έχει κάθε κράτος να το κάνει. Κάτι το οποίο επίσης ανέφερε ο κύριος ε, Μποργέτζο σήμερα το πρωί είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη σύγκρουση των συμφερόντων. Ποιος εκδίδει αυτούς τους τίτλους, ποιος τους αξιολογεί, ποιος ε, δρά ως ενδιάμεσος μεταξύ των ε, μέσων και της αγοράς και ποιος συμβουλεύει τους επενδυτές οι σύμβουλοι. Αυτοί όλοι πρέπει να είναι διαφορετικά υποκείμενα. Δεν μπορεί το ίδιο υποκείμενο να κάνει ταυτόχρονα τις ίδιες δουλειές. Κυρίως όσον αφορά τις, ε, τους οίκους αξιολόγησης που συγχωρήστε με, δεν είναι μια στήρα επίθεση αυτή. Ε, ήταν πάρα πολύ κακή η διαχείριση που έκανα στην κατάσταση, αρκεί να δούμε τα τριπλά α, τα τρία α που δίνονταν σε επιχειρήσεις που κάποιες μέρες μετά χρεοκοπούσαν. Εγώ νομίζω ότι η αξιολόγηση, το να ε, κάποιο, αξιολογεί κάποιο τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και αυτού που τα εκδίδουν, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δημοσίου συμφέροντο. Επομένω, θα πρέπει να γίνεται από δημόσιου φορεί. Είτε είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή ή το σύστημα, και εδώ συμφωνώ μαζί σας κυρία Μπερές, να είναι οι κεντρικές τράπεζες κάθε χώρας μέλους. Και εδώ θα ήθελα να το προσθέσω αυτό ε, στην άποψή σας με την οποία συμφωνώ. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε και τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Ε, τις ανεξάρτητες αρχές του χρηματιστηρίου, για τις χρηματοοικονομικές αγορές, για τις ασφαλιστικές αγορές, οι οποίες πρέπει να είναι αυστηρές και αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να επιμολύνονται από την εισαγωγή μεταβλητών που έχουν προκύψει από τις πολιτικές εξουσίες. Θα πρέπει να αποτελούνται από υψηλά εστάμενους ε, με πολύ καλά προσόντα που δεν θα τους έχουν προτείνει λόμπι ε, ε, για συγκεκριμένες πιέσεις. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Εμείς έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν αρκεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε ίσως μια οικονομική και μια χρηματοοικονομική κοινή πολιτική. Δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν περιορίζεται στο ρόλο του συντονιστή των πολιτικών ε, της κάθε χώρας μέλους, αλλά έχει τη δική της πολιτική και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τη φορολογική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε οι, αυτοί οι οποίοι θα συλλέγουμε τους φόρους, οι φορείς πράκτορε. Απλώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ομαλοποιήσουμε τις ε, διάφορες φορολογικές διαφορές, όπως για παράδειγμα τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και αυτή την ε, ανταγωνιστικότητα που υπάρχει ε, στους φόρους για να μπορεί κάποιος να ε, προσελκύει εισοδήματα και κεφάλαια. Ένα τελευταίο στοιχείο για τη διακυβέρνηση. Απολογιστικής πλευράς αυτή τη φορά. διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια τάση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσουν την τέταρτη και την έβδομη οδηγία ε, σε θέματα επιχειρήσεων. Από ένα ε, σύστημα το οποίο ήταν πολύ προληπτικό που καθόριζε ε, ποια ήταν τα εισοδήματα μιας επιχείρησης βάσει ενός ιστορικού κόστους, περάσαμε σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στο μέλλον. Εκεί λοιπόν που λειτουργούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι διαφορές που αξιολογούνται, όχι οι συναλλαγές οι οποίες έγιναν, αλλά και η βάση που χρησιμοποιείται και το πώς μοιράζονται τα έσοδα στους μετόχους ε, υπό τη μορφή μερισμάτων. Αυτά για την τροποποίηση που συζητάτε για την τέταρτη οδηγία είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τους κανόνες της διακυβέρνησης τώρα, πολύ σύντομα. Εμείς έχουμε διαχειριστές και διευθύνοντες σύμβουλες, συμβούλους επιχειρήσεων που δρούν για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αποζημιώνονται για αυτές τις πολύ σύντομες ε, προοπτικές. Ε, κατά την άποψή μου θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το θέμα. Η, είτε η διακυβέρνηση της επιχείρησης, είτε οι αποζημιώσεις, τα ποσά τα οποία λαμβάνουν ε, οι μάνατζερ σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ε, ε, ένα πιο μακρόπνο σχέδιο, να είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμα, να μην ε, προσφέρεται ως πάροχος υπηρεσιών αυτός που ελέγχει τις ίδιες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ως επιχειρηματική σύμβουλη ή ως φορολογική σύμβουλη. Θα πρέπει ε, εντό των επιχειρήσεων να μην υπάρχει καμία σύγκρουση, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα σύγκρουση συμφερόντων. Και κάτι τελευταίο, και με αυτό ολοκληρώνω, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο επεσήμανα ως τελευταίο σημείο του εγγράφου μου και που πραγματικά έλαβα και υπόψη στο σχέδιο, ε, λαμβάνεται συγγνώμη υπόψη στο σχέδιο έκθεσης κυρίας ε, Περές. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε στη διοίκηση μιας επιχείρησης όλους αυτούς που συμμετέχουν στην εργασία μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να ε, υλοποιήσουμε ένα σύστημα σαν το σύστημα το οποίο υπάρχει στην ομοθέσια της Γερμανίας. Και στο σύστημα αυτό οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα ε, εποπτείας. Για παράδειγμα, στην Άωση Στάτη και σε άλλους αντίστοιχους οργανισμούς. Σήμερα το πρωί ε, άκουσα στη σημερινή συνεδρίαση έναν Ευρωβουλευτή, ο οποίος δεν είναι μόνο από τη χώρα μου, αλλά είναι και από την πόλη μου, είναι από τη ε, Τζένοβα, τον κύριο Κοφεράτη, ο οποίος ε, είπε ότι τον ανησυχεί αυτό το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων. Το κατανοώ. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό από τους εργοδότες ε, διότι έλεγαν ότι αν συμμετέχουν στα κέρδη, ποιο θα συμμετέχει στις απώλειες και στις ζημίες. Υπάρχει ένα άρθρο στη, και στη μεταπολεμική περίοδο αλλά και στην ε, δεκαετία του 70. Εάν τα συνδικάτα είχαν εκπροσώπηση από άνθρωπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, με ποιον θα είχαν γίνει πάλι των τάξεων. νομίζω ότι αυτή η λύση είναι μία από τις πολλές λύσεις που δεν θα επιτρέψουν στο κεφάλαιο να ε, υπησέρχεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διότι ε, από την κρίση της εργασίας πλήττονται και το κεφάλαιο αλλά και οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον τρίτο ομιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Θα προσπαθήσω να περιορίσω τα σχόλιά μου σε πιο πρακτικά θέματα, σε γενικά σχόλια. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε την έκθεση αυτή. Είναι γεμάτη από πολύ καλές ιδέες, ιδίως αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα όραμα. Ε, αντιμετωπίζουμε μια σειρά κρίσεων χωρίς πολιτικές πρωτοβουλίες για να δούμε τι θα γίνει και ό,τι γίνεται ανταποκρίνεται σε κάτι που έχει γίνει, δεν υπάρχει μία πρωτοβουλία πουθενά. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι παρόλο που επρόκειτο για μία σειρά και συλλογή πολλών διαφερουσών ιδεών, έχει ενωθεί σε αυτό το κείμενο κατά τέτοιο τρόπο που όταν το διαβάσει κανένας δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Θα ωφελούνται σημαντικά όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλεται για να συμβάλλεται στην έλλειψη ιδεών και πολιτικών πρωτοβουλειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είχε δοθεί μια τέτοια δομή που ή θα υπήρχαν κάποιες βασικές αρχές ή μηνύματα, μηχανισμοί συνοχής και συνέχισης, ούτω ώστε κάποιο που το διαβάζει να πει Α, αυτό θα πρέπει να γίνει. Και εκτό αυτού να, έχει η δυνατότητα το κοινοβούλιο να καταλάβει ότι ωραία, μα ζητάνε να κάνουν κάποια πράγματα και υπάρχουν μηχανισμοί για να ακολουθήσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή για τίποτα άλλο παρά το να υπάρχει ένα πολιτικό όραμα που λείπει αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την εντολή της Επιτροπής Κρίσης που διαφέρει από τη δική σας ίσως, είναι ότι είχε την εντολή να έχει μια πιο οριστική προσέγγιση, καθολική αντιμετώπιση και όχι να επιστρέψει στις λεπτομέρειες. Θα ήταν καλό ίσως να μπορέσουμε να σωματώσουμε τα διάφορα, α, τις διάφορες στοιχές. Οι προσπάθειες για την ε, ενσωμάτωση των κοινωνικών και των οικονομικών τυχών ίσως είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Επιτροπή Κρίσης έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει και το βραχυπρόθεσμο και το μακρυπρόθεσμο. Ναι, η σημερινή κρίση ξεκίνησε από προβλήματα subprime. Είναι κάτι που ακολουθείται τώρα από μια κοινωνική επίσης κρίση, αλλά τα προβλήματα στην Ευρώπη <laughs> χρονολογούνται από πολύ πιο παλιά. Να πούμε ότι ναι, το άμεσο κόστος ήταν πάρα πολύ ψηλό, το φορολογικό κόστος ήταν πάρα πολύ ψηλό. Αλλά το κύριο πρόβλημα ήταν η μη σωστή κατανομή των πόρων εδώ και δύο και τρει δεκαετίες. Γιατί το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έκανε ό,τι πρέπει να κάνει και η οικονομική διακυβέρνηση δεν ε, ήταν αυτή που έπρεπε. Μακροπρόθεσμη ανεργία, διαφορετικά προβλήματα κλπ. λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν καλό λοιπόν η έκθεση να μην εξετάσει βραχυπρόθεσμα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και τα κοινωνικά θέματα. Το καλύτερο θα ήταν να υπάρχουν κάποια κύρια πολιτικά μηνύματα προς το Συμβούλιο, προς την Κομισιόν, προς τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Επίσης θα ήταν όμως μια πλούσια πηγή ιδεών για πολιτική. Μια στιγμή κατά την οποία τα περισσότερα ε, Υπουργεία Οικονομικών δεν ξέρουν ακριβώ τι να κάνουν, εσεί καταβάλλετε μεγάλε προσπάθειε, είχατε διάφορε ακροάσει και πρέπει τώρα να πείτε τι πρέπει να γίνει. Θα ήταν λοιπόν καλό να έχετε έτσι ορισμένες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται επίσης να ολοκληρωθεί το κενό που υπάρχει στη λειτουργία, δηλαδή τα άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα όπως εσείς. Χρειάζονται λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό όργανο όπως εσείς να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Στη ΣΥΠΑ ε, υπάρχει η Επιτροπή Κρίσης η οποία είχε ακρόασεις για να δει τι θα γίνει για να την εντόπιση κρίση κρίσης και μαθαίνει πώς θα μπορέσει να προχωρήσει. Η Υποεπιτροπή Ερευνών της Γερουσίας έχει κάνει ακροάσεις για το Lehman Brothers και το Goldman Sachs αλλά δεν ξέρω κατά πόσον για την ε, Deutsche Bank ή άλλες έχουμε κάτι ε, παρόμοιο. Δηλαδή ε, στην Ευρώπη το θέμα του, του προς ποιον υπάρχει ανάγκη ε, να είναι υπολογή, το τι έχει γίνει με όλες αυτές τις δέσμες για τη διάσωση των τραπεζών κλπ. Δεν είναι καθόλου σαφές. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι η Deutsche Bank διαφέρει και τόσο πολύ από την Goldman Sachs. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τούτο λεχθέντος, οι σημαντικές μικροοικονομικέ πληκτές είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο έχει κάποια κινητικότητα, κεφαλαίου κλπ. Αλλά δεν υπάρχει φορολογικό συντονισμό. οι αγορέ απασχόληση είναι κατακαιρμασμένε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ή μπορούμε να επανέλθουμε στο να είμαστε μεμονωμένα κράτη-μέλη ή μπορούμε να προχωρήσουμε προς κάτι που είναι μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση. Η μπορουμε να προχωρησουμε προ κατι είναι ενωση εμει βρισκομαστε στη μεση αβέβαια προ τα που θα κλείνουμε. Και γι' αυτό η συζήτηση για περισσότερη φορολογική συντονιστική προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή ή χρειαζόμαστε πλήρη Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν χρειαζόμαστε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μισό από αυτό και μισό από το άλλο δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. ό,τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν στην προπόθεση ότι θα υπάρχει σημαντική σύγκληση. Ξέρουμε ότι αυτό δεν έγινε. Και για λόγους πολιτιστικών διαφορών διαφορών ε, διαστρωτικών της οικονομίας για διάφορους διάφορους λόγους. Αυτό που θα πρέπει να δούμε τώρα είναι πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα ότι θα έχουμε αποκλίνωση στις εθνικές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και η πρόκληση είναι ακριβώς πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό χωρίς να οδηγηθούμε σε μια ασταθή κατάσταση. Γενικά, το μήνυμά μου θα ήταν ότι χρειάζεται να αυξηθεί ο χώρος των πολιτικών. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορες κρίσεις ε, περιβαλλοντολογικές, ε, απασχόλησης, ε, χρηματοπιστωτικές, κοινωνικές και δεν έχουμε ακόμα τα μέσα πολιτικής ούτε στο εθνικό επίπεδο, αλλά ιδίω όχι στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι προκλήσει. Ακόμα και αν δούμε αυτό που λένε πολλοί πολλοί Υπουργοί Οικονομικών ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μέσο πολιτική για να αντιμετωπιστεί ε, κάθε πρόβλημα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε με ένα μέσο να αντιμετωπιστούμε πολλά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν έχουν αρκετά μέσα πολιτικά. Παραδείγματο χάρη. Θα μπορούμε πολλά να μάθουμε τι αντισόμενε χώρε. Γιατί τι είχαμε. Είχαμε μια αντικατάσταση στην Ευρώπη. Και εγκαταλείψαμε διάφορα μέσο πολιτικών που είχαμε υπήρχαν, ε, ε, ε, υπάρχουν δυνατότητες διάσωσης, υπήρχαν κεφάλια αποθηματικού κλπ. που τα εγκαταλείψαμε και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα πολύ πιο σημαντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολύ σημαντικότερη κρίση απασχόλησης από ό,τι έχουμε εμείς. για μας αυτά είναι καινούρια σε άλλες χώρες τα είχαν πολλά χρόνια. Πολλά μαθήματα μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από τις χώρες αυτές. Τι θα κάνουμε με το πλάνο, πώς θα αναδιορθώσουμε, πώς θα έχουμε περισσότερα όργανα της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο από θέματα ε, δανείων κλπ. Και, και μια διαστατική πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει ευέλικτα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις σημερινές προκλήσεις αλλά και καινούριε προκλήσεις που θα μας παρουσιαστούν. Αυτό θα ήταν το κύριο μου μήνυμα. Όσον αφορά ποιε είναι οι ιδέες με τις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να δούμε βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τώρα την ύφαση. Δεν θέλουμε να κατακαιρματιστεί η Ευρωζώνη. Σημαντικό αυτό. Θέλουμε να ελεγχιστοποιήσουμε ε, τα πλήγματα στην κοινωνική δυχή. Ε, κάποιες ιδέες έτσι, θα σας τα δώσω γραπτά αν θέλετε, ορισμένα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι προβληματικές οι ροές των δανείων, γιατί οι τράπεζες έχουν ε, αυτή τη στιγμή ωφέλη, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν και μερίσματα. Παραδείγματο χάρη, ένα πανευρωπαϊκό μορατόριο για την πληρωμή ε, υπερβολικών αμοιβών. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε τι θα γίνει με τις αποφάσεις που βασίζονται στη Συμφωνία της Βασιλείας. Δηλαδή, η επιδότηση που δίνει στις τράπεζες στο χαμηλό επιτόκιο αυτή τη στιγμή δεν πάει στις τσέπες των, ε, ε, των επενδυτών ή των μετόχων, αλλά στην επαναφορά της εμπιστοσύνης. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους καλούς φόρους, τους φόρους της ακτακτικότητας ή φόρους για ε, βιομηχανίες που μολύνουν υπερβολικά. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε την ανάγκη περισσότερων φορολογικών εισόδων, αλλά ε, φορολογικών εισόδων που δεν θα πλήξουν τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με μια σειρά κινήσεων καλά μελετημένων κατά της φοροδιαφυγής. Ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά χρειάζεται να γίνουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ένωσης. Υπάρχουν επίσης ε, ανάγκη μεσοπρόθεσμα μέτρα, παραδείγματο χάρη. Οι ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις να είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες των ε, χρηματοδοτικών συστημάτων. Γιατί ένα από τα προβλήματα είναι ότι κάθε νομοθεσία που προτείνεται αυτή είναι μια νομοθεσία αντίδρασης. Κανένας δεν αναρωτιέται ποιο είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρειαζόμαστε, ποιο είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα υποστηρίξει την ε, ανάπτυξη που χρειαζόμαστε για να έχουμε τα συστήματα που χρειαζόμαστε και τι σημαίνει αυτό για την ρυθμιστική συζήτηση που γίνεται άλλες ενδιαφέρουσες ε, ιδέες, ε, ε, μετοχές που σχετίζονται με το ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε την κατάσταση κρίσης, το βλέπουμε αυτό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι και, και προσεχώς θα έχουμε κάθε είδους κρίσης και θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους που έχουν απομείνει να σχολιάσουν. Και να αρχίσω με εσάς, Περβάνς, που είσαστε η συγγήτρια. Για την πληροφορία σας, εδώ στο πάνελ, έχω να πω ότι είχαμε μια συζήτηση. Ο καθηγητής Διάντζελος ήταν εδώ για την έκθεση αυτή, αλλά τώρα μας παρουσιάσετε οπωσδήποτε νέες σκέψεις. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ στην κοινοβουλευτική εργασία υπάρχουν ορισμένα άχαρα πράγματα και δύσκολα, άρατα, όπου άλλα βέμα που έχουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να προχωρήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν που συμβάλλατε σε αυτά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια πρωτόγονη αν θέλετε μέθοδο γιατί έχω καταγράψει όλες τις ε, παρατηρήσεις που είχα για να συμβάλλω πολιτικά αν θέλετε. Όσον αφορά το να δούμε ποια είναι τα διακυβεύματα των λόγων ε, και των αιτιών της κρίσης, αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο τεχνικό. Εγώ όταν ίσως κάπως προκλητικά είχα ξεκινήσει με την πρώτη γραμμή της έκθεσης, είχα πει ότι ο πρώτος λόγος της κρίσης ήταν η ανισότητα κατανομής των εισόδων. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επίπτωση της κρίσης. Η κρίση βέβαια καταστά ακόμα πιο σοβαρά τα προβλήματα αυτά της διαφοράς της ε, κατανομής των εισόδων. Αλλά κατά την προέλευση της ε, κρίσης, στην πηγή της κρίσης, το θέμα της ανισότητας των εισόδων και της ανισότητας κατανομής θέμενες αξίες είναι τμήμα από τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα του κεφαλαίου και πιο μικρή κινητικότητα της εργασίας. Αλλά αυτά πάντως είναι στοιχεία που δεν είναι επιπτώσεις αλλά είναι αιτίες κατά κάποιο τρόπο της κρίσης. σε αυτά που είπε και ο κ. Κάμπος δεν κατάλαβα αν είπατε ότι η θεσμική διαδικασία είναι καλή ή όχι καλή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας δυναμισμός και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το θεσμικό τρίγωνο όσον αφορά τον ευρωπαϊκό δυναμισμό έχει οπωσδήποτε πολλά πλεονεκτήματα. Και όταν δω την ομάδα εργασία τη οποία προεδρεύει ο πρόεδρο Σέμα Φαν έχω να πω ότι εκεί υπάρχει κάτι το οποίο με ανησυχεί. Δηλαδή, ή θα πρέπει να παραμείνουμε στο, στην κατάσταση της σημερινής διακυβέρνησης της ζώνης ευρώ ή ότι θα πρέπει οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων να κατευθύνουν τη ευρωζώνη. Όχι, όχι. Η πρόταση που κάνω στην παράγραφο 154 που είναι μια πρόταση θεσμικής εξέλιξης είναι κατά τη γνώμη πάρα σημαντική. Γιατί αυτό είναι το μέσο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που έχουμε από τότε που περάσαμε στην Ευρωζώνη, δηλαδή να συνδυάσουμε τις ικανότητες της ε, Κομισιόν και την ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας τον εθνικό χαρακτήρα των φορολογικών και οικονομικών πολιτικών. Ειλικρινά, πιστεύω ότι όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής και Νομισματικής ε, ε, Ένωσης υπάρχουν δύο πράγματα. Ή χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε κανόνες πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήταν επαρκής μέχρι στιγμή και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτή την πτυχή μέχρι σκασμού και ότι αυτή η πειθαρχία θα επιτρέψει κάποια στιγμή σε αυτό το μεγάλο οικονομικό χώρο που είναι η Ευρωζώνη να είναι ανταγωνιστική σε διεθνέ επίπεδο κλπ. Εγώ, εγώ προφανώ δεν το πιστεύω, αλλά είναι και αυτό μια δυνατότητα, ένα δυνατό σενάριο. Το άλλο είναι να θεωρήσουμε ότι μια ολοκληρωμένη νομισματική ζώνη θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένο προπολογισμό, ολοκληρωμένη οικονομία και θα πρέπει σύμφωνα με το μοντέλο των Αμερικανών να έχουμε ένα προπολογισμό του 20% θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά όχι μεσοπρόθεσμα. Ας μην κλείσουμε την πόρτα σε αυτή την άγουσα. Ας ήμουν όμως ρεαλιστές. Να μην ζητάμε το αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια γράφη το πρωί. Μεταξύ των δύο αυτών, χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη αυτό που ξέρουμε σήμερα, ότι η αποστάσεις ανταγωνιστότητας είναι τεράστιες, επιδεινώθηκαν από τότε που περάσαμε στο ευρώ και γι' αυτό η ιδέα ότι ο καθένας, και αυτό είναι το μέλλον της έκθεσης, ο καθένας να πρέπει να τακτοποιήσει τα του οίκου του, δεν αρκεί για να καταλήξουμε σε μια πραγματική διακυβέρνηση, οικονομική διακυβέρνηση του, της Ευρωζώνης, όπως τη χρειαζόμαστε. Είπατε κύριε Κάμπος, ότι η έκθεση προσανατολίζεται στην ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, ναι, φυσικό είναι. Ε, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό είναι ακριβώς η ιδιαιτερότητα της έκθεσης. Ότι εκτός από τις, από τις ε, ε προτάσεις κομισιών που καθορίζονται λίγο πολύ από ό,τι πρότεινε πρόκειται να δείξουν τα κρατημέλη και τι σκέφτονται τα κρατημέλη. Εδώ, σε αυτό το σώμα, έχουμε δυνατότητα να έχουμε ένα όραμα τη ευρωπαϊκή διάσταση, άσχετα από τι θα κάνει κάθε κυβέρνηση. Ο καθένα πρέπει να κάνει δουλειά του, βέβαια. Όσον αφορά τη φορολογική εναρμόνιση. Χαίρομαι που ζώστε την άποψή μου. Όσον αφορά το μισθούς, δύο θέματα. Εγώ δεν προτείνω εναρμόνιση του ελαχίστου μισθού, γιατί πρέπει να ξεχνάμε το αρχικό κείμενο ήταν το γαλλικό. Το γαλλικό κείμενο δεν αναφέρεται σε εναρμόνιση των μισθών, αναφέρεται όχι στον ελάχιστο μισθό, το πρωτότυπο, αλλά στο ελάχιστο εισόδημα. Και δεύτερον, εγώ δεν μιλάω για εναρμόνιση, αλλά για ορισμό σε κάθε χώρα μέλος ενός ελαχίστου ε, εισοδήματος συγγνώμη, ανάλογο με τις προϋποθέσεις της κάθε χώρας. Όσον αφορά την αποταμίευση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, βέβαια στην έκθεση αναφέρεται πολύ το θέμα του αμερικανικού θέματος, γιατί σε διεθνή κλίμακα ήταν αυτό ένα σημαντικό σημείο, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές είχαμε την τάση να ε, μην ανησυχούμε και πολύ για την αύξηση του δανεισμού των οικοκυριών. Συμπληρωμένο και μεγάλων δυσκολών για ορισμένου από εμά που θέλαμε να καταδικάσουμε τα κυλιόμενα αυτά δάνεια και ήρθαν κάποιοι και μας είπανε μα αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή καινοτομία οικονομική και δεν πρέπει να την ε, κατηγορήσετε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω το θέμα του, ε, της χρέωσης και της υπερχρέωσης των νοικοκυριών είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και από την άλλη μεριά, οι παραδόσεις αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι επίσης σημαντικοί. Κύριε Ντιάγγελης, ε, σας ευχαριστώ πολύ για όσα αναφέρατε όσον αφορά το φόρο για τις ε, επιχειρήσεις ή για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, είναι πράγματα τα οποία δεν συμφωνούμε. Όσον αφορά όμως το θέμα του boycott της Goldman Sachs, σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Είναι ίσως μια πρόταση η οποία κάνει ορισμένου να χαμογελούν, να αισθάνονται του έχει προκαλέσει κάτι. Ε, ένα περιφερειακό συμβούλιο της Γαλλίας χθες αποφάσισε ένα μποϊκότ όλων εκείνων των τραπεζών που έχουν επενδύσει στους φορολογικούς παραδείσους. Αυτή η προσέγγιση δεν αρκεί να κατηγορεί κανένας, αλλά όσον αφορά τις ε, αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις υπάρχει ε, κάποια κάποιο συσχετισμό με τα μέσα που χρησιμοποιούν, εκεί είναι σημαντικό. Τώρα θα μου πείτε, γιατί την Goldman Sachs και όχι άλλου. Ε, είναι προφανέ. Γιατί η Goldman Sachs εκπροσωπεί την πιο επιτυχή επιχείρηση σε αυτό το τομέα γιατί ο κύκλος εργασιών ε, διπλασιάστηκε. Απ' την άλλη μεριά όμως, και νομίζω ότι συμφωνούμε πάνω σε αυτό, όσον αφορά τους παράγοντες εκκίνησης της κρίσης, το θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας και το θέμα που ανέφερε ο κύριος Καπούρ της αποσύνδεσης των ε, χρηματοδοτικών μηχανισμών και των πραγματικών αναγκών δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και ούτε μπορούμε να παραβλέψουμε το ρόλο εκείνων των, των οργανώσεων που πραγματικά ενστενήθηκαν πλήρες αυτό το επιχειρησιακό μοντέλο. Ξέρω από αυτά που άκουσα για τη Γαλλία, ορισμένοι στην αγορά σήμερα προτιμούν πραγματικά άλλε ε, τράπεζες επενδύσεων, άλλε δομέ επενδύσεων και όχι την Goldman Sachs. Λοιπόν, εάν οι άμεση ενδιαφερόμενοι αναρωτιούνται τι γίνεται με το θέμα, θα πρέπει να το κάνουν και πολιτικά υπεύθυνοι. Ε, θα πρέπει τώρα να δούμε κατά πόσο πρέπει να, να έχουμε μια διεθνή διακυβέρνηση ή όχι δεν θέλω να πούμε ότι εμείς είμαστε ένα όργανο που είναι αρμόδιο για τα πάντα, αλλά είπα και το έχουν εξετάσει με τον ε, πρόεδρο στην προηγούμενη θητεία προσεκτικά αυτό το θέμα. Αν κοιτάξω τα πρότυπα λογιστικής ή την Επιτροπή της Βασιλείας. Εκεί υπάρχει ένας αυτοέλεγχος γιατί κατηγορήθηκε το επιχειρησιακό του ε, μοντέλο και υπάρχει τώρα μια ομάδα ε, ελέγχου, επιθεώρησης, μονιτόρνη που τους ελέγχει αυτούς τους, τους λογιστές που κάνουν τους ελέγχους. Εγώ είχα πει ότι θα, πρέπει να ε, εξαρτηθεί από το ε, FMI, e, από το Διεθνές Μονιτομισμικό Ταμείο. Το θέμα του πού υπάρχει αναφορά για να βγει ο καθένα από τον κέτο του, ούτως ώστε τα λογιστικά αυτά πρότυπα να μην προετοιμάζονται από τους ίδιους αυτούς τους επιθεωρητές λογιστές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τι ανάγκε της ε, χρηματοπιστικής σταθερότητας, γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο της κρίσης. Και έτσι που είναι πολύπλοκο ο κόσμος σήμερα, ε, ο καθένα μπήκε στο δικό του γκέτο και έκανε το δικό του ό,τι ήθελε εκεί. Γιατί ξεχνάμε ότι είναι λογιστικό πρότυπο δεν είναι ένας αριθμός. Μπορεί να έχει και έναν ε, οικονομικό δυναμισμό. Άμα εσείς επικρίνετε την δίκαια αξία, την fair value, προφανώς, προφανώς οι επιθεωρητές είναι εκείνοι που δεν θα το έχουν ίσως κατά νου θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι ασυχέ μα να έχουμε καλύτερη ισορροπία. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, βαθμολόγηση, νομίζω υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία στην έκθεση. Όταν στην τελευταία θητεία είχαμε τη συζήτηση για τι υπηρεσίες αυτή τη βαθμολόγηση, ετέχει το θέμα κατά πόσον όταν βαθμολογείται μία έκδοση μετοχών από κάποια ε, επιχείρηση. Ή έχουμε τη βαθμολόγηση των ε, χρεών κλπ. Και για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντος, δεν ξέρω, μήπως θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε το μοντέλο αυτό της επιχείρησης. Αυτή η βαθμολόγηση να γίνεται δηλαδή από τον επενδυτή. Είναι μια συζήτηση που ξεκινάει τώρα. Απλώ σα δείχνω την ιδέα αυτή Έχουμε και του δύο ομολόγου στο, στο Κογκρέσο και διάβασα μόλι τώρα τα πρακτικά μια ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή τη οποία προεδρεύει ο κύριος Άγγελης. Δηλαδή που υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε δηλώσει πάνω στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται το τριπλό α για κάποια προϊόντα κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σόνικα Πόρ για όσα μας είπε. Δεν, έχουμε δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Έχουμε πραγματικά μια οριστική εντολή. Έτσι την ορίσαμε. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, πώς θα διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. για να τελειοποιήσουμε την έκθεση. Όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής ε, Επιτροπής, ε, νομίζω ότι αναφέρθηκα προηγουμένως όταν απάντησα στον κύριο Κάμπος για τα τρία δυνατά πρότυπα, όπου φτάνουμε σε αυτή την ιδέα που θα έχουμε κάτι παραπάνω, που θα έχουμε κάτι λιγότερο. Το status quo βέβαια δεν επιτρέπεται. Και μετά η ιδέα ότι χρειάζεται διακασμασμό που έχει κατά νου τι ανάγκε τη οικονομία. ε, αυτό είναι ένα τμήμα των ανησυχιών μα και ελπίζω ότι πραγματικά διατυπώνεται αρκετά έντονα στην έκθεση και υπάρχει σε κάποια, ε, σε κάποια παράγραφο που δεν θυμάμαι ακριβώ τον αριθμό τη, αλλά αναφέρεται ρητά. σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, η, Thank you Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία και για την ενθαρρυντική συζήτηση. Θεωρείτε ότι αυτή η κρίση είναι μια ε, κρίση των οικονομικών, της οικονομικής επιστήμης δηλαδή, της επιστήμης των οικονομικών. Ένας καθηγητής οικονομικών στη Φιλανδία αναφέρθηκε στα αποτελέσματα μιας έρευνας που ανελήφθη πριν από την ε, έκρηξη της κρίσης και μας είπε ότι όσο, πιο, ε, όσο περισσότερο σπουδάζει κανείς οικονομικά, τόσο πιο αδυσόπιτος γίνεται. Και αυτό ισχύει γιατί μία πλευρά της εκπαίδευσης βασίζεται σε ε, μαθηματικά στοιχεία με σενάρια απόλυτου κέρδους ή απόλυτης ζημίας. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευση, το σύστημα παιδείας έτσι ώστε να εμπεριέχει και ένα σύστημα αξιών, έτσι ώστε ο καθένας να καταλαβαίνει τις επιπτώσεις των, ε, των διαφόρων οικονομικών σχημάτων. Θα ήθελα και ο κύριος Μποργέζιο να παρέμβει και μετά να επανέλθετε εσείς στα τρία σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για αυτή την περαιτέρω συνεισφορά άκρος ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές. Ε, σε σχέση με την, ε, το έγγραφο που οδήγησε σε μια συγκεκριμένη συζήτηση δηλαδή και στην απότοκη συζήτηση. Ίσως ε, δεν κατάλαβα εγώ κάτι καλά ή δόθηκαν διευκρινήσεις ως προς τις ενδείξεις, περαιτέρω ενδείξεις που θα έπρεπε να διασαφινιστούν. Ε, ως προς την έκθεση του κυρίου Ντεάντζελης, ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να χτίσουμε ένα συνικό τείχος ως προς τη διαφοροποίηση που γίνεται αυτή ε, ως προς τα συμφέροντα ή αυτό το παιχνίδι ρόλων ε, στον τομέα της διαμεσολάβησης στα χρηματοπιστωτικά. Υπάρχει μεγάλη ρήξη συμφερόντων και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνηση, δηλαδή αυτή η επιθετική στάση που θα πρέπει να καταδείξει κανείς για να υπερασπιστεί είτε το κεφάλαιο είτε τους αποταμιευτές. Νομίζω ότι στην ε, επικείμενη συζήτηση δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη μία ενδεχόμενη κοινή απόφαση για τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί οι φούσκες συνεχώς υπάρχουν και υπάρχουν και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Άρα στην τελική έκθεση δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο των ε, Ιδρυμάτων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας των οργανισμών αυτών. Θα πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Δεν θα πρέπει να ακολουθούμε μία ε, πολιτική που να διέπεται μόνο από πολιτικούς. Θα πρέπει να δούμε πώς έχουν και οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη μελλοντική μας οικονομική πορεία. Δηλαδή να δούμε και τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων πολιτών. Και εν τέλει, ως προς προτάσεις της έκθεσης για την συμμετοχή των εργαζομένων, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς για το ποια είναι τα εμπόδια σε αυτή την πορεία. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν εμπόδια για αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία είναι αναγκαία, διότι εκεί που διεξήχθη καλός, κατέδειξε το γεγονός ότι υπηρετεί μια σύγχρονη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθετε στα ερωτήματα οι τρεις συνάδελφοι. Μπορείτε να αρχίσετε εσείς κύριε Κάμπος. Πέντε λεπτά εντάξει. Ναι, μπορείτε να έχετε 5 λεπτά, 5-6 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Uh, just, um, on... Σε σχέση με ορισμένα σχόλια που κατέγραψα, συμφωνώ ότι θα πρέπει, συμφωνώ, θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με τα θεσμικά μέσα που διαθέτουμε. Νομίζω ότι η εξισορρόπηση εξουσιών μεταξύ θερμικών οργάνων, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών ε, πρόκειται για μια ε, μεταβατική πορεία η οποία είναι μεταβατική. Και βεβαίως η ανταπόκρισή μας το δείχνει αυτό. Δεν θα ήθελα να επικρίνω το έγγραφο. Θα ήθελα απλώς να πω ότι το έγγραφο αυτό ε, δείχνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερος επιμερισμός εξουσιών στο φορολογικό τομέα. Διάβασα το ε, αγγλικό κείμενο, το κείμενο στα αγγλικά Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι κατά πόσο ο ελάχιστος μισθός έχει επίπτωση στην απασχολησιμότητα. Θα πρέπει να είμαστε ε, πάρα πολύ σαφείς ως προς τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πρότασης και βεβαίως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Με απασχολεί λοιπόν αυτό το θέμα διότι ε, ε, υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς το μισθολογικό που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ε, χαίρομαι που συμφωνείτε ότι το αποταμιευτικό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και ότι είναι δύσκολο δεν, πρέπει, ότι δεν, πρέπει, σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί. Ως το θέμα της εκπαίδευσης της οικονομικές σπουδές, ε, εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν θεωρώ ότι είμαι αδυσόπιτο στην προσέγγιση μου. Αυτό το λέω στη χώρα μου πολλές φορές και στην τηλεόραση γίνονται συζητήσεις για την κρίση και είχα τονίσει αρκετές φορές και έλαβα πολλά ε, email που με συνεχάρισαν. Δηλαδή, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, θα πρέπει να... ότι τα οικονομικά ναι μεν διέπονται και έχουν ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, αλλά όταν σπούδασα εγώ οικονομικά, για ένα χρόνο, τον πρώτο χρόνο σπουδάζαμε και φιλοσοφία. Τώρα είναι επιλογή δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, βασικές φιλοσοφικές αρχές δεν διδάσκονται πια στις οικονομικές σπουδές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κανένας είναι αδίστακτος επειδή σπουδάζει οικονομικά. Ασχολούμαι, έχω ένα μάθημα την διεθνή οικονομία, χρηματοοικονομικά ε, και είναι διαφορετικοί οι φοιτητέ μου. Ήδη από 18-19 χρονών οι φοιτητέ μου έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Το καταλαβαίνω από τις ερωτήσεις που υποβάλλουν, από τον τρόπο σκέψης τους δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό σε αυτό που, το, που διδάσκουμε, γιατί εμεί το ίδιο διδάσκουμε. Απλώ πρόκειται για διαφορετικού ανθρώπου. Δεν λέω ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι χειρότερο, απλώ οι άνθρωποι διαφέρουν και πριν αρχίσουν σπουδέ. Τα μαθηματικά είναι μία γλώσσα, όπως τα αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά. αλλά δεν είναι τόσο λαμπερές γλώσσες, δεν μπορούμε να γράψουμε ποίηση με τα μαθηματικά. Είναι μια αυστηρή γλώσσα, δεν κάνουμε λογικά λάθη χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά. Δηλαδή αν τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται καλώς, ε, καλώς έχουν. Τα μαθηματικά πρότυπα βοηθούν τους ανθρώπους. Δεν είναι υποκατάστατα σκέψεις, αλλά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πολλά ζητήματα. Και πολύ συχνά οι φοιτητέ εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτά τα πρότυπα σαν να ήταν πραγματικότητα. Ένα πρότυπο είναι μια καλή μίμηση της πραγματικότητας, στην καλύτερη περίπτωση. Και δεν είμαι ο μόνος που διδάσκει τους φοιτητές κατά αυτόν τον τρόπο αλλά όταν διδάσκονται και ορισμένες βασικές αρχές της φιλοσοφίας θα βοηθούσε ιδιαίτερα και όχι μόνο στα μαθηματικά. Καταρχάς, μια πολύ σύντομη απάντηση, δεν πρόκειται βέβαια για απάντηση, προς την κυρία Γιακονσάρη. Ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρα το όνομά σας σωστά. Οι οικονομολόγοι. Εγώ διδάσκω σε ένα τμήμα οικονομικών, διδάσκω εμπορικό δίκαιο και πάντα λέω στους συναδέλφους, αν ένας γιατρός κάνει λάθος σε μία επέμβαση, πληρώνει διότι έχει ευθύνη. Αν ένας δικηγόρος χάσει μια υπόθεση, στη χειρότερη περίπτωση θα χάσει τον ε, πελάτη του. Οι επιχειρήσεις, οι λογιστές, αν κάνουν λάθος, πρέπει να καταβάλουν ε, τεράστια ποσά αν χρεοκοπήσει η επιχείρησή τους. Έχετε δει ποτέ οικονομολόγο να του επιρρύπτονται ευθύνε αν κάνει λάθος οι οικονομολόγοι με κάθε σεβασμό και φιλία που τρέφω προς αυτό μπορούν να πούνε «Α, κάναμε λάθος τις πράξεις» ή ε, «Σωστά ήταν εμένα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, άλλαξαν τα πράγματα και δεν έχουμε καμία ευθύνη». Γι' αυτό λοιπόν για τις υποθέσεις των οικονομολόγων να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Δεύτερον, κύριε Μπερές, εγώ σας ευχαριστώ διότι κυρίως τα σημεία τα οποία σας επεσήμενα εγώ για την ε, έκθεσή σας, εκφράζοντας μεν τη διαφωνία μου, αλλά είναι τέσσερα και μόνο σημεία στα 200 ε, τα οποία διαφωνώ. Επομένως θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η απάντησή σας, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν με έπεισε, αλλά θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση για τη φορολογική πολιτική. Εγώ μιλούσα για φορολογική ομοιομορφία, όχι για τα ελάχιστα εισοδήματα, αλλά για φορολογική ομοιομορφία, κυρίως όσον αφορά στον εταιρικό φόρο, δηλαδή φορολογία στα εισοδήματα μιας επιχείρησης και κυρίως ε, φορολογία κεφαλαίου, στα εισοδήματα κεφαλαίου, διότι αν η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και ούτω καθεξής ε, έχουν ανταγωνισμό μεταξύ των απλώς και μόνο για να προσελκύουν περισσότερα κεφάλαια, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτε με, αυτή, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει να δράσει δια της βίας με την πυθό είτε με άλλους μέσους, ώστε, με άλλα μέσα, συγγνώμη, ώστε τα εισοδήματα να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο για να υπάρχει ομοιομορφία μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών και να μπορούμε να έχουμε ελευθερία μετακίνησης ε, ανθρώπων, κεφαλαίων και επιχειρήσεων. Τελεία. Κύριε Μποργέτσιο, ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων νομίζω ότι τα έχω πει όλα και κάτι επιπλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αρχές που σας ε, ανέφερα, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλα τα ισχυρά λόμπι του τραπεζικού κόσμου. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ρίξουμε και εμείς μία ε, πέτρα, να δούμε μακροπρόθεσμα ε, τι αποτέλεσμα θα έχει στο βάλτο. Ως προς το θέμα της συμμετοχής. Ένα πράγμα μόνο να πω. Δυστυχώς λόγω περιορισμένου χρόνου χρειάστηκα να περιορίσω την παρέμβασή μου και ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής. Σκεφτείτε τη Γερμανία. Μια Γερμανία που βγαίνει από τον πόλεμο το 1945 κατεστραμμένη, όπως και η Ιταλία άλλωστε. Το γεγονός ότι μπορεί η Γερμανία να σηκώσει κεφάλι και να γίνει η οικονομική δύναμη που είναι αυτή τη στιγμή, οφείλεται κατά βάση, κατά την άποψή μου, στα βασικά κίνητρα που έχει, στις επιχειρήσεις. Το να υπάρχει διάλογος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο από τις πολιτικές αρχές και από τον νομοθέτη. Η υποχρέωση λοιπόν να υπάρχει διάλογος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας και εργαζομένων δηλαδή, Γι' αυτό και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Κοφεράτη, το συμπατριώτη μου, που είμαστε από την ίδια πόλη. Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση, πρέπει να υπάρχει διάλογος. Και ο σωστός χώρος για το διάλογο είναι στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι, άλλα φόρα για τις συλλογικέ συμβάσεις και το καθεξής. Αλλά στις επιχειρήσεις είναι να υπάρχει ένα συμβούλιο επιτήρησης, ένα σύστχατ, ένα κονσέγγι ένα surveillance ένα ανώτατο όργανο το οποίο θα εποπτεύει. Δεν δίνονται εκτελεστικές αποφάσεις, δίνονται κατευθύνσεις προς τις επιχειρήσεις. Αλλιώς το μόνο που θα έχουμε ε, είναι ότι θα έχουμε μια συνεχή αντιπαράθεση και όποιος δεν πλήρωσε δεν θα πληρώσει ούτε και τώρα. Ο Σόνι Δεν μελέτησα οικονομικά, δεν σπούδασα οικονομικά, αλλά ορισμένες φορές διδάσκω οικονομικά. κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Πρώτον, τα οικονομικά που μαθαίνουμε. Και εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν φτάσει κάποιος στο μάστερ ή στο διδακτορικό του, πρέπει να ξεχάσει όλα όσα έχει μάθει στα οικονομικά στο πρώτο έτος. Όλα αυτά θα πρέπει να του έχουν γίνει δεύτερη φύση στο μεταξύ. Όλες οι έννοιες που μαθαίνονται στο πρώτο έτος στα οικονομικά πρέπει να μαθευτούν εκεί γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να κάνεις καμία δουλειά ή ε, δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στο διδακτορικό σου. Εάν κάποιος λοιπόν ασχολείται συνεχώς με το όλο φάσμα των οικονομικών, τα οποία έχουν ξεκινήσει με υποθέσεις που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα έχουμε υποθέσεις οι οποίες μπαίνουν ακριβώς στο μυαλό μας και γίνονται μνήμη. Και εδώ έρχεται και αυτό το παράδειγμα που ακούσαμε με τη μελέτη φιλοσοφίας. Οι οικονομολόγοι λοιπόν δεν θα πρέπει να μελετούν μόνο οικονομικά, θα πρέπει να σπουδάζουν και φιλοσοφία και άλλα μαθήματα ώστε να μπορούν να έχουν μια ευρύτερη προοπτική. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η φυσική περιβάλλοντος. αυτή έχει επισέλθει σε πολλά οικονομικά μοντέλα και σε πολλά χρηματοπιστωτικά μοντέλα. Όπως έλεγε και ο Κέινς, έχει Λάθο και μάλιστα αυτό είναι ακριβέ. Δηλαδή αυτό που ήθελε να πει είναι ότι είναι καλύτερο να κάνει κάποιο λάθο, από το να μην είναι, και να είναι βέβαιο ότι είναι λάθο αυτό που κάνει, από το να μην είναι ε, ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Τα οικονομικά μοντέλα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο ρόλο για τον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν υπάρχει χρηματοοικονομικός τομέα στα μοντέλα οικονομικών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα να μας πούνε για το τι ακριβώς κάνουμε σε περίπτωση κρίσης. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Εγώ ήμουνα στην ε, εναρκτήρια συνεδρίαση ε, του συνεδρίου για το Economic Thinking. Ε, κάποιοι οικονομολόγοι το έκαναν αυτό μαζί με τον George Soros και θα πρέπει να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν όμως αυτό που μας μένει είναι τα οικονομικά του πρώτου έτους. Για να επανέλθω τώρα στην Goldman Sachs, εγώ ήμουνα ε, σύμβουλος στρατηγικής ε, στην κυβέρνηση πριν από κάποια χρόνια και όταν συζητούσαμε τα θέματα των οικονομικών παραδείσων, των φορολογικών παραδείσων, υπήρχαν αρκετά συμβούλια που είχαν αναλάβει κάποια μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι δημόσιες ε, συμβάσεις μόνο για όσους δεν ε, έχουν δουλειές με φορολογικούς παραδείσους. Και το θέμα με την Goldman Sachs είναι ότι είτε θα καθορίσουμε μια σειρά από κριτήρια και θα λέμε ότι κάποια τράπεζα που δεν έχει επιδοτήσει και δεν έχει φορολογικού παραδόσεις ή δεν ε, έχει νομικέ εκκρεμότητε ή οποιαδήποτε τράπεζα ε, έχει αποδείξει ότι δεν είναι συνένοχο στο έγκλημα κλπ. Ε, πρέπει να υπάρχουν κάπου κάποια κριτήρια. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή είναι ότι υπάρχει αυτός ο μύθος της Goldman Sachs. Η κρίση έχει προκαλέσει ένα μύθο ότι η Goldman Sachs κάπου διαφέρει από τις υπόλοιπες. Εάν είχαμε κρίση και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε γλιτώσει τους πάντες, η Goldman Sachs θα είχε αποτύχει όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει αυτός ο, ο μύθος της Goldman Sachs. Είναι απλώς ο τρόπος που, που ε, έδρασε η ιστορία. Αν είχαν πάει αλλιώς τα πράγματα, ε, θα ήταν άλλη. Η Morgan Stanley, π.χ. μπορεί να είχε περισσότερα έσοδα κάπου δημιουργήθηκε η λανθασμένη εντύπωση ότι οι τράπεζες διαφέρουν μεταξύ τους και ότι η Goldman Sachs είναι η μόνη η οποία μπόρεσε να γλιτώσει από το σκάνδαλο με τα subprimes, με τα ανυπόθηκα δάνεια και ε, διατηρείται, συντηρείται αυτός ο μύχο της Goldman Sachs και αυτό είναι κρίμα γιατί μπορεί να δημιουργήσει και σε διάφορα, ε, σε λανθασμένα ε, συμπεράσματα πολιτική. Μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, οι Barclays, οι UBS και όλες οι γερμανικές τράπεζες, η Deutsche Bank, είναι κατά κάποιο τρόπο καλύτερες ή διαφορετικές ή δεν έχουν συμμετάσχει τόσο πολύ στο έγκλημα. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι έτσι. Και αυτό που είναι πιο τρομακτικό σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, συζητώνται αυτά τα πράγματα, συγκρούσεις συμφορέων με την Goldman Sachs και πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν, τα λόμπι, όλα αυτά γίνονται υπογείως στην Ευρώπη και κλεισμένων των θυρών και δεν υπάρχει καμία σοβαρή συζήτηση για τράπεζες, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ μεγάλες για να ε, αποτύχουν. Στην Ευρώπη υπάρχει 200 με 300% ε, των εσόδων ε, των τραπεζών που είναι άνω του ΑΕΠ μιας χώρας. Ε, αυτές οι τράπεζες δεν έχουν την πολυτέλεια να αποτύχουν. δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα μόνο της Goldman Sachs. Η Deutsche το έκανε αυτό και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο και έχει πείσει τους πάντες ότι η Goldman Sachs είναι μόνη προβληματική. Δεν είναι αλήθεια. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό ε, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ε, Είναι μια ε, επιχείρηση που έχει εκπροσώπους ορκωτών λογιστών και εκεί λέγεται ότι οτιδήποτε έχει τέτοιο βαθμό δημόσια σημασία θα πρέπει να ελέγχεται και θα πρέπει να υπάρχει μια κυβερνητική δομή που θα ελέγχει κάτι αντίστοιχο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, ή τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης υπάρχει το θέμα της άνησης κατανομής. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι κάτι το οποίο αναφέρεται μεν στην έκθεση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το επισημάνουμε ακόμα περισσότερο. Το γεγονό ότι έχουμε δύο ίδιοι ανθρώπου στην κοινωνία. Ανθρώπου σαν εσά και εμένα, που το μεγαλύτερο μέρο του εισοδήματό μα προκύπτει από μισθού. και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν εισοδήματα και ακίνητα και ε, κερδίζουν τα περισσότερα εισοδήματά του από εκεί. Και το θέμα είναι ότι η ανισότητα αυτή σε κάποιο βαθμό έχει προκύψει και από την ε, ε, υπερβολική πίστοση. Έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα από τις πιστώσεις για παράδειγμα, διότι οι άνθρωποι σαν εμένα και εσά που δεν έχουν εισοδήματα από αυτά, έχουν μόνο από τους μισθούς, έχουν πλέον μεγάλη διαφορά στα εισοδήματά τους με τους ανθρώπους που είναι εισοδηματίες. Αυτός που έβγαζε 5 δολάρια θα βγάζει 55 δολάρια. Ε, κάποιος ο οποίος έχει ε, πάρα πολλά έσοδα ε, θα ξοδέψει ουσιαστικά ποσά σαν να ξοδεύαμε εμείς 2 δολάρια, διότι πόσα μπορεί να ξοδέψει πια κάποιος. Αν ξυπνήσετε αύριο το πρωί, δεν θα σας το συστήνω αυτό, αλλά αν ξυπνήσετε αύριο το πρωί και ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο, όπου έχει γίνει αναδιανομή του κόστους με πιο ισότιμο τρόπο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, θα έχετε ένα πολύ ε, μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικής αύξησης και μεγαλύτερη ε, αύξηση στη ζήτηση. Δεν συστήνω να γίνει αυτό. Σχόλιο εκτό μικροφώνου από τον πρόεδρο. Ίσως σα το συστήνω, τέλος πάντων. Αλλά να σας πω δύο πράγματα εδώ. Μας ανησυχούσαν ήδη πάρα πολύ οι μεγάλες ανισότητες ε, και λόγω των δημοσιονομικών προοπτικών. Κάποια τμήματα της κοινωνίας ενδιαφέρονται για τα οικονομικά, κάποια άλλη όχι. Υπήρχε όμω και το γεγονό ότι δεν υπήρχε συσσωρευμένη ζήτηση. Αυτό που έκανε η κρίση ήταν ότι έχει ε, δημιουργήσει ένα τρίτο πολύ σημαντικό λόγο από πολιτική σκοπιά για την ανισότητα. Και είναι το γεγονό ότι τα μεγάλα ποσοστά ανισότητα δημιουργούν ε, μεγάλο πληθωρισμό στι τιμέ των και αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ε, θα οδηγήσει πάντα σε κατάρρευση και σε οικονομική κρίση σαν αυτή που έχουμε. Και αυτή η πτυχή δεν έχει συζητηθεί επαρκώ. Πλέον λοιπόν έχουμε τρεις λόγους για την αντιμετώπιση της ανισότητας και όχι δύο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω κάποια πράγματα από την ε, πείρα μου για το συνικό τείχος. Τα συνικά τείχη δεν δουλεύουν, ε, είναι, δεν λειτουργούν, είναι διαβρωτά. Έχετε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικούς ε, ορόφους, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση και άμα του πείτε ότι μπορούν να αυξήσουν τα εισοδήματά του κατά 20-30% θα κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Ήμουνα στη Lehman Brothers πριν από 8-9 χρόνια και την πρώτη εβδομάδα που ήμουν εκεί είδα τους τρεις ε, τέσσερις από, τους διάσημα, τα τρία, διάσημα σημικά τείχη να καταραίουν. Και αυτό είναι αυτό το οποίο γίνεται καθημερινώς. Και έτσι θα έχει κατάσταση. Αυτό είχαμε στην Ευρώπη και τώρα όλο ένα και περισσότερο και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το γεγονό ότι αυξάνει συνεχώς και ε, το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σημαίνει ότι έχουμε χρήματα από απλού ανθρώπους, σαν εσά και εμένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για περισσότερε επενδύσει κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εμεί έχουμε επενδύσει χρήματα στι τράπεζε πιστεύαμε ότι θα είναι πιο υπεύθυνοι, θα μας τα φυλάνε, θα μας τα κρατάνε ασφαλή έχουν, αλλά δεν έκαναν αυτό το πράγμα οι τράπεζες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το δυνατικό διαχωρισμό των διαφορετικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι πολύ πιο προχωρημένη συζήτηση αυτή στι ΗΠΑ. Στην Ευρώπη δυστυχώ δεν συζητάται ακόμα. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δούμε και το θέμα τη ποικιλομορφία πολύ μικρές τράπεζες, ε, είδαμε για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιες τοπικές τράπεζες που έχουν προβλήματα. Είναι εκτεθειμένες σε μεγάλους παραγοντές κινδύνου στην τοπική κοινωνία. Εάν για παράδειγμα κλείσει μια επιχείρηση ή ένα εργοστάσιο σε, μια, σε ένα μικρό μέρος, η τράπεζα που χρηματοδοτεί όλους τους εργαζομένους ε, της, του εργοστασίου θα κλείσει και αυτή. η πραγματική ποικιλομορφία προκύπτει σε μεσαίο επίπεδο, διότι και οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Όταν είσαι μεσαίο μεγέθης, είσαι εκτεθειμένος σε δύο ή τρεις πόλεις, δεν έχεις όμως πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και δεν... Ε, ε, είναι μια πολύ μεγάλη μοιρασιά, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καλάθι που πρέπει να τα βάλεις όλα και εδώ δημιουργούνται προβλήματα. Μια τελευταία παρατήρηση. Η αναλογία κινδύνου τη σύγκρουση συμφερόντων. Ένα συνάδελφό μου λέει ότι θα πουλούσε τη μάνα του για 10 εκατομμύρια δολάρια. Εγώ δεν θα την πουλούσα τη μάνα μου, αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι άλλο παπαδαγγέλιο. Όταν λοιπόν συζητούμε τέτοια πράγματα και λέει ότι κάποιο μπορεί να πάρει χρήματα για κάτι, μπορεί κάποιο να σκότωνε άνθρωπο για 10.000 δολάρια, για 20.000 δολάρια. Άνθρωποι, λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν φρικτά πράγματα για πάρα πολύ μικρά ποσά. Εάν λοιπόν κάποιο ανταμείβει μία συμπεριφορά που δεν ε, θεωρείται παράνομη στην κοινωνία και δεν ε, κάποιο να πληρώσει κάποιο τίμημα, ε, συ, μου λέτε ότι εγώ δεν θα το κάνω, είναι απαράδεκτο. Αν είναι κάποιο πολύ καλό οδοντίατρο, μπορεί να δουλεύει 18 ώρε τη μέρα, μπορεί να βγάζει 1000 ευρώ την ημέρα, αλλά δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 18.000 ευρώ την ημέρα. Αν είσαι τραπεζίτης, κάνει μια συμφωνία που σου ε, αποφέρει κέρδος 100 εκατομμύρια ευρώ, είναι μια συμφωνία ή 100.000 δολάρια και είναι ε, ε, μια συμφωνία ενός εκατομμυρίου δολαρίων και αν αλλάξει, βάλεις ένα μηδενικό, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Είναι δικά σου χρήματα, δεν δικά μου και πληρώνεσαι 10 φορές περισσότερο από ό,τι θα πληρωνώσουν. Και ε, σου λέει κανεί ότι θα πει όχι και δεν θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια στα τραπεζικά συστήματα και η απόδοση είναι πολύ πιο ασθενή από ό,τι σε άλλα συστήματα. Και ε, τα σωστά οικονομικά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αντικατοπτρίζουν αυτό όλο. Ευχαριστώ. Βάτε τα ακουστικά και θα μιλήσω γερμανικά παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τρεις ε, εδώ στο, κυρίους εδώ στο πάνελ για τις συμβολές τους και γραπτά και προφορικά και την απάντηση των ερωτήσεων και των σχολείων. Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω σαν σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, ένα σχόλιο. Δεν είναι κανένα αντίθετο με μοντέλα ή με πρότυπα. Μοντέλο είναι χρήσιμο. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο τα μοντέλα αυτά να κυριαρχούν τη διαδικασία και κατά κάποιο τρόπο να ανεξαρτοποιηθούν και να οδηγήσουν στο σοκ που είδαμε τελευταία, όταν ε, έπεσαν τα χρηματιστήρια κατά χίλιους πόντους γιατί υπήρχε κάποιο μοντέλο που κινεί το αυτόματα κλπ. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται ας πούμε. Ο Κέινς εκφράστηκε με σαφήνεια, με κατανόηση. Δεν χρειαζόταν ε, σελίδες επί σελίδων μαθηματικών μοντέλων. Και ένας τέος φοιτητή ε, μετά πέντε χρόνια που θα γίνει από το Μεσημπέ, όλα αυτά τα που δεν τα κατάλαβε. Κατάλαβε που ανέφερε ο κύριος Ντάντζελε. Έχετε δίκιο ότι η ε, τελευταία αναλύση Ποιο θα πληρώσει, εσείς και εγώ, ο κατανοητής. Εάν όμω μιλάμε για έναν φόρο για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι 0,05 και 0,03% της συναλλαγής. Οπότε δεν παίζει ρόλο, γιατί αν σκεφτείτε ότι η τράπεζα ζητάει 0,5 και 1% για μια συναλλαγή, τίποτα δεν είναι λοιπόν το 0,05. Αν όμω το συλλέξουμε, το συναθρήσουμε, το ποσό είναι τεράστιο. Εγώ όπω φιλελεύθερο είμαι ούτως άλλως κατά των φορολογικών αυξήσεων συνήθω. εγώ δεν έχω να πω αυτά που θα φανταζόστε ότι θα έλεγα. Δεν έχω αυτές τις επιφυλάξεις που φανταζόμαστε. Όσον αφορά το κύριο Σόνι Καπούρ και την επαναδιανομή του ισοδύναμα, θα σας πω κάτι από τη χώρα μου όπου έχουμε μοσπαρκά κρατήδια και ξέρετε ορισμένα οι χαρακτήρια έχουν έλλειμμα, ορισμένα βρίσκονται καλύτερη θέση και οι πλούσιοι επιδοτούν τους φτωχούς. Υπάρχει μια ανακατανομή των ισοδυναμάτων. Δυστυχώς εκείνα τα κράτη που χρόνο με χρόνο χρηματοδοτούνται δεν ξεπέρασαν ποτέ την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται γιατί δεν έχουν κανένα, ε, κανένα και μάλιστα εκείνες οι χώρες, που, εκείνα τα κρατήρια, συγγνώμη, πολλές φορές που επιδοτούν τα άλλα, στο τέλος βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από εκείνα τα οποία έχουν υποδοτήσει. Ε, δεν είναι πράγματα αυτά. Επίσης είπατε, κύριε Καπούρ, είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο φορολογικά έσοδα. Ωραία είναι πάντα περισσότερα φορολογικά έσοδα, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ και 30 χρόνια, εκτός από το τελευταίο έτος, είχαμε συνεχώς περισσότερα φορολογικά έσοδα στη χώρα μου. Παρόλο όμως την αύξηση των κρατικών εσόδων, είχαμε ε, πολύ μεγαλύτερη αύξηση των δαπανών. Δηλαδή μόλις ανακαλύπτουμε ε, μια νέα πηγή εσόδου, ξέρω εγώ, για το διοξείδιο του άνθρακα ή για το περιβάλλον ή κάτι τέτοιο, εκείνη τη στιγμή αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι δαπάνες μας. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο για αποταμίευση. Ερωτήσεις τώρα. Πρώτον, ο καθένας παρακαλώ να κάνετε τρεις συγκεκριμένες δηλώσεις κλειδί σε σχέση με την κρίση. Ποιες θα ήταν αυτές οι τρεις ο καθένας. Δεύτερον, θεωρείτε ότι όσον αφορά τη Βασιλεία και στην G20 που προετοιμάζουν προτάσεις που δεν έχουν όμως δεσμευτικό χαρακτήρα, Πιστεύετε πρέπει να αποχωρήσουμε λίγο και να δώσουμε σε αυτά έναν ε, χαρακτήρα σύμβασης για να δεσμευτικά και μετά όταν περάσω στις ε, υπηρεσίες αξιολόγηση των δανείων εκείνες πάντα λένε μα εμείς μόνο γνωμοδοτούμε. Δεν είναι τίποτα δεσμευτικό αυτό που λέμε. Μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε ένα βήμα και να πούμε εσείς είσαστε υπεύθυνοι για αυτό που μας λέτε. Δεν είναι μόνο γνωμοδότηση, γιατί έτσι πάνω σε τη βάση αυτών που λέτε βλαμβάνω πάρα πολύ σημαντικέ αποφάσει. Θα ήθελα να πάω λίγο πίσω σε αυτό το παράδειγμα που αναφέρθηκε για την επαναδιανομή του εισοδήματος και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οπωσδήποτε ε, κάτι τέτοιο θα αύξηνε την κατανάλωση και αυτό θα προωθούσε την ανάπτυξη φέτος και του χρόνου. Αλλά δεν θα υπάρχει όμως μια πραγματική τάση ανάπτυξης, γιατί μια αύξηση της κατανάλωτης θα σήμαινε μείωση του ποσοστού αποτεμίευσης. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, η αναδιανομή του εισοδήματος από τη μια στιγμή στην άλλη θα αύξηνε την κατανάλωση, αλλά δεν θα οδηγούσε σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Όσον αφορά τα μαθηματικά μοντέλα το έγγραφο αναφέρεται συχνά σε μαθηματικά πρότυπα. Αν πρόκειται για οικονομικά ή χρηματοπιστωτικά, θα συμφωνούσα. Αλλά τα μαθηματικά δεν είναι αυτό που είναι το σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τα μοντέλα αυτά. Εγώ έχω πάει σε διάφορα θεσμικά όργανα και έχω ρωτήσει, ας πούμε, 2,3 δεν μπορεί να είναι το σωστό αριθμητικό στοιχείο για του χρόνου. Και η απάντηση είναι ναι, μα το μοντέλο μας τόσο βγάζει. Μα δεν είναι καλή αυτή η απάντηση. Ένα μοντέλο πρόκειται να βοηθήσει. Πρέπει κανένας να είναι προσεκτικός. Εάν το μοντέλο οδηγεί σε, ε, σε κακές απαντήσεις, αυτό οφείλεται στο ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι το σωστό, δεν είναι καλό. Δεν είναι λοιπόν κάτι που αντικαθιστά τις σκέψεις μας το μοντέλο. Η κυρία Περές ε, διακόπτη. Κοιτάξτε, Εάν πάτε στην παράγραφο 114, δεν αναφέρεται στα πρότυπα, αλλά στη χρήση των μοντέλων. Η θεωρία του σημερινή πλήση θα μπορούσε να ξαναθέσει αμφισβήτη τον τρόπο χρησιμοποίηση ορισμένων μαθηματικών μοντέλων. Ακριβώ αυτό που λέτε και εσεί, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έλεγα ότι αν λέγατε όχι μαθηματικά αλλά χρηματοπιστωτικά θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας. Στην οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν θαυμάσια μοντέλα και τους ε, και κάνουν, δίνουν την εντύπωση ότι ε, εκεί πρέπει να βαστούν. Λένε, ας πούμε, ο κίνδυνος είναι 7,2. Ναι, μα δεν είναι ο κίνδυνος 7,2. Αυτό είναι μία μέθοδος ε, να μετρηθεί κατά κάποιον τρόπο πολύ χοντρικά ο κίνδυνος. Ο φόρος Τέρμπιν. Θαυμάσια ιδέα. Γιατί κατά βάση δεν έχει επίπτωση στις μακροπρόθεσμες συναλλαγές αν πάει από τη μια χώρα στην άλλη 10 εκατομμύρια σήμερα και σε 10 χρόνια τα ξανά επαναφέρω, αυτό δεν μετράει. Δεν είναι μηδέν. Άμα το κάνω αυτό όμως κάθε ώρα, ε, τότε βέβαια είναι σημαντικό. Δηλαδή, και επιβάλλει Ρώσεις στις βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές κινήσεις χωρίς να επιβάλλει καιρώσει στις μακροπρόθεσμες πραγματικές κινήσεις κεφαλαίου. Είναι καλή ιδέα. Αυτό που λένε οι χρηματοπιστικοί κύκλοι είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Όλοι καταλαβαίνουν όμως ότι η ιδέα του τόρμπινταξ ε, του φόρου Τόρμπιν, είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως βέβαια ρίξει λίγο άμμο στους καλά λαδωμένες ε, στα καλά ρωτωμένα γρανάζια της ε, οικονομίας και θα ήταν καλό αυτό. Θα ήταν καλό εάν οι, ε, οι υπηρεσίες αξιολόγησης ήταν αγκασμένες να αιτιολογήσουν αυτό που λέει. Πρόσφατα το rating της Πορτογαλίας μειώθηκε. Και δεν υπήρχε καμία αιτιολόγηση. Δεν υπήρχε καμία αλλαγή εδώ και έξι μήνες ή μήνες ή ένα χρόνο. κινείται η αγορά προς κάποια εσφαλμένη κατεύθυνση. Ίσως καμιά φορά γίνεται αυτό και για καλούς λόγους και όχι κακούς. Αλλά δεν υπήρχε καμία δικαιολογία, καμία αιτιολόγηση. Αν λοιπόν είναι αναγκασμένοι πλήρως να αιτιολογούν την απόφασή τους, θα ήταν πολύ πιο προσεκτική στην βαθμολόγηση αυτή που κάνουν, στο writing. Κάτι άλλο. Όταν υπάρχουν κανονισμοί, παραδείγματο χάρη ότι η βαθμολόγηση κράτους δεν μπορεί να αλλάξει πιο συχνά παρά μια φορά το χρόνο προ δύο κατευθύνσει, και προ τα πάνω και προ τα κάτω. Τότε θα είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί θα ξέρουν ότι αυτή η θεφανολογία που θα δώσουν σήμερα θα πρέπει να την κρατήσουν ένα χρόνο. Και δεν θα ακολουθούν κάποιε μόδε χρηματοστοπιστικών αγορών, θα πρέπει να κάνουν μια πραγματική αξιολόγηση του κράτου. Υπάρχουν λοιπόν πολλά μικρά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για να αυξηθεί η αξιοπιστία των υπηρεσιών αυτών αξιολόγηση rating agencies. Υπάρχει βέβαια μεγάλη ε, σύγκρουση φερόντα μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και των τραπεζών που τους αναθέτουν κλπ. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν το θέμα. Αλλά σου ακούσετε κάποιες ιδέες σχετικά. Αυτά είχα να πω πρόεδρε. Τα, οι, κύριες, οι τρεις ε, κύριες βασικές ιδέες δεν μας τις είπατε. Ως προς τα πρότυπα, τα οικονομετρικά, οικονομικών και μαθηματικών συνάμα. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσω. Νομίζω ότι η κυρία Μπερές έχει δίκιο όταν λέει ότι το πρότυπο καθ' αυτό είναι ουδέτερο. Θα πρέπει να δούμε τι χρήση θα γίνει για να δούμε τι επιπτώσεις απορρέουν από το πρότυπο. Αυτό που είδαμε είναι ότι στις τράπεζες τα πρότυπα α, άλλαξαν την πείρα των πεπειραμένων ε, τραπεζιτών που βρίσκονται στην αγορά πάρα πολλά χρόνια. Άρα η, πείρα τους είναι καλύτερη από τα πρότυπα, αλλά δυστυχώς ακολουθούν πρότυπα, μαθηματικά πρότυπα και όχι την πείρα τους. Συμφωνώ μαζί σας υπό την έννοια ότι οι αξιολογήσεις που εξαρτώνται από την πείρα μπορούν να αλλάξουν πολύ πιο άμεσα από αυτές που βασίζονται σε αυστηρά πρότυπα, αυστηρά σταθερά πρότυπα. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν. Τα πρότυπα είναι συλλογιστικοί μηχανισμοί που πολλές φορές εάν δεν προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα δεδομένα δίνουν μια άλλη εικόνα από αυτή της πραγματικότητας. Δεν είμαι βεβαίως ο καταλληλότερος να δώσω μια απάντηση σε αντίθεση με τους συναδέλφους για την επανακατανομή των εισοδημάτων. Αυτό είναι έργο των κρατών αυτή τη στιγμή που απορρέει από μια φορολογική πολιτική. Άρα, ή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάσουν σε μια συμφωνία για να, ε, δώσουν στην, να προσδώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος της ε, φορολογικής πολιτικής, όπως είπα πριν. Μίλησα για τον φόρο των επιχειρήσεων, των ε, κεφαλαιουχικών αγαθών, αλλά το θέμα δεν βρίσκεται εδώ το θέμα τίθεται σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, ελπίζοντας να είναι αρκετά συνετά να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Όσο προς τους οργανισμούς αξιολόγησης ε, πιστοληπτικής ικανότητας, ε, είπατε ότι βρίσκονται πίσω από συγκεκριμένα χαρακόμματα, αλλά ε, πολλές φορές η γνωμοδότηση δεν οδηγεί και σε ευθύνες αλλά πάμε λίγο σε βάθος. Αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τις αγορές. Ή από την πλευρά της προστασίας και των αποταμιευτών και των επενδυτών. Ποιος πληρώνει τώρα αυτούς τους οργανισμούς. Αυτούς τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας, γιατί είναι μια επιχείρηση είναι ένα, ένα εμπόριο, είναι μια εταιρεία. Τι αποκομίζουν από αυτό. Ξέρουμε ποια είναι τα έξοδά τους, τα έξοδα προσωπικού, τα ε, πρότυπα που αγοράζουν από εξειδικευμένους οργανισμούς, από το σύστημα ε, πληροφορικής, αλλά το, το, το κέρδος τους ποιο είναι διότι οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι όπως τα χρηματιστήρια, τα οποία ε, ε, ε, στην ουσία πληρώνονται από τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για να εποπτεύουν αυτή τη δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δηλαδή πληρώνονται από τις τράπεζες. Τώρα, από τα έσοδα των οργανισμών αυτών, ένα μέρος των εσόδων μπορεί να αφορά και προβλέψεις χρήσης χρηματοοικονομικών μοντέλων. Άρα, πώς γίνεται η διαβούλευση για, για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά όργανα τα οποία μετά θα πρέπει να αξιολογήσουν. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι τι αντίκτυπος υπάρχει ως προς το ρόλο τους, ας το πούμε, και ως προς τι επίπτωση έχουν. Έτσι τουλάχιστον κινείται η έκθεση Μπερές, δηλαδή η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να γίνει μόνο από αυτούς τους οργανισμούς που έχουν έναν δημόσιο ρόλο. Πώς τώρα αξιολογούν. Αξιολογούν χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δημόσια ή ιδιωτικά και σε αυτούς που εκδίδουν χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κράτη, ε, ε, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Εάν πρόκειται τώρα για κεντρικές ε, τράπεζες ε, ορισμένων κρατών, δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα προϊόντα που εκδίδουν τα ίδια τα κράτη, ας πούμε τα ομόλογα. Εκεί χρειάζεται αποκλειστική, υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Όμως μπορούν να αξιολογήσουν, δηλαδή να βαθμολογήσουν τα προϊόντα ή τις αρχές έκδοσης προϊόντων του, της χρηματο, χρηματοπιστωτικής αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ε, εμβαθύνουμε το όλο θέμα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δημοσιοποιηθεί αυτή η λειτουργία rating αξιολόγησης. Let me start with your last question first, which are the key... Ως προς το τελευταίο που ρωτήσατε, ποια είναι τα βασικά στοιχεία εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα στοιχεία και όχι τρία. Το πρώτο είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλαπλά μέτρα Άρα υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επέκταση μέσων σε επίπεδο κεντρικών, ας πούμε, τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της αξιολόγησης τραπεζών κλπ. Το δεύτερο είναι ότι η συζήτηση για την κρίση αφορά περισσότερο τη ρύθμιση, αλλά σημασία έχει πώς έχει η ροή, διότι το νερό πέφτει από το βουνό κάτω στο λόφο, στις υπόρειες του λόφου και στο τέλος στην ε, θάλασσα. Άρα τα κέρδη ορίζονται από τη ρύθμιση. Η ρύθμιση λέει αυτό μπορείτε να κάνετε, εκείνο δεν μπορείτε να το κάνετε. Πέρα από αυτό, όμως, αυτό που έχει σημασία είναι η φορολόγηση, τα equity, τα περιθώρια μόχλευσης, οι μακροχρόνιες συναλλαγές, οι οποίες φορολογούνται ή δεν φορολογούνται, ποια είναι η κεφαλαιοχική απόδοση και ούτω καθεξής. Και βεβαίως και η νομισματική πολιτική, δηλαδή προληπτικά μέσα, prudential, που ορίζουν και τα επιτόκια. Άρα αυτό που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι ένα σύστημα και να δείτε πού διασταυρώνονται αυτά τα τρία στοιχεία. Δηλαδή πού περνά αυτή η ροή, η χρηματοπιστωτική ροή. Χρειαζόσαστε έξυπνα ρυθμιστικά, φορολογικά μέτρα που να ε, συμπνέουν, να έχουν μια σύμπνοια. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν όλα έχουν καλώς, τότε αυτό ίδιο ισχύει και για τις ε, πολιτικές και για τις χρηματοπιστωτικές ροές. Δεν είμαστε έτοιμοι για αντιμετώπιση κατάστασης κρίσης. Άρα χρειάζεται να αποδώσουμε μεγαλύτερη πρόσοχη. Δηλαδή όπως ζητάμε από τις τράπεζες να κάνουν δοκιμές, να δουν τι θα γίνει με ενδυνάμει αποτυχίες, ενδυνάμει ζημίες, ενδυνάμει αστάθειες και να χτίσουν αναχώματα, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την αιγίδα της Κομισιόν ή ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Χρειαζόμαστε υποχρεωτικό προγραμματισμό, δεσμευτικό προγραμματισμό και πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να κινηθούμε. Γιατί μιλάμε για το πού πήγαμε, τι δεν πήγε καλά και πώς μπορούμε να τα παλώσουμε. Θα πρέπει να έχουμε ολιστική προσέγγιση στα ειδικότερα σημεία. Ως προς το, τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και σε σχέση με αυτά που είπε η Bundesbank δεν θα πρέπει να είναι ενιαίος ο φόρος, αλλά διάφοροι δίκτες, διάφορα ποσοστά που να ισχύουν ας πούμε για την αγορά παραγόγων. Άλλο η αγορά παραγόγων και άλλο η αγορά του χρηματιστηρίου. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Δεύτερον, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Βραζιλία και η Ινδία χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που μας δίνουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα για να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα του δημοσίου χρέους καλύτερα. Αλλά δεν έχουμε παρκείς πληροφορίες για τον όγκο των συναλλαγών. Άρα αυτό είναι πρόσθετο μέσο. Πληροφορίες. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, που είναι οι συναλλαγές στον κυβερνοχώρο, δεν διέπονταν από κάτι, δεν ξέραμε ποιος ε, συναλλασσόταν με ποιον, ποιο ήταν το αντίπαλο δέος και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μια ηχνηλάτηση των συναλλαγών και έτσι μπορούμε να φορολογήσουμε και ανάλογα. Έτσι βλέπουμε ποιες είναι οι ρυθμιστικές αλλαγές που επέρχονται και το άλλο αντιστάθμισμα είναι ότι οι ρυθμιστικές αλλαγές ως προς τα παράγωγα μας οδηγούν στο να μπορούμε να φορολογήσουμε καλύτερα τις συναλλαγές. Αυτό λέει και η βιομηχανία συναλλαγών. Σε ορισμένες αγορές είναι ήδη εύκολο, θα γίνει ακόμα πιο εύκολο και σε άλλες αλλαγές, ιδιαίτερα ως προς τα παράγωγα, ως προς τον συστημικό κίνδυνο. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό, αυτή είναι η ρύθμιση. Εμείς τι κάνουμε, οι ΜΜΕ δανείζονται από τράπεζες. Οι πολυεθνικές πάνε στην κεφαλουχική αγορά. Άρα η αγορά και οι τράπεζες είναι δύο διαφορετικές πτυχές του χρηματοπιστωτικού. Συζητάμε βεβαίως και τον φόρο των τραπεζών που αφορούν τους ισολογισμούς των τραπεζών καθαρά. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη κερδοφορία που πάει στην αγορά και στο τέλος ο φόρος καταβάλλεται από τους μικρομεσαίους. Άρα πρόκειται για ένα συμπληρωματικό σχήμα φορολόγησης, να φορολογήσουμε τα hedge funds, την χρηματοπιστωτική αγορά και όχι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. θα πρέπει να πρόκειται για δύο συμπληρωματικά σχήματα ρύθμισης. Μιλάμε για κεφαλουχικές ανάγκες για να σταθεροποιήσουμε τις τράπεζες. Δεν υπάρχει όμως μια κυκλική πορεία που να διέπει τις αγορές. Άρα το να επιβάλλουμε ένα φόρο όπως κάνει η Κίνα όπου αυξάνουμε το ποσοστό όταν υπερθερμαίνεται η αγορά, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα κυκλικά φαινόμενα. Και επίσης μπορούμε να έχουμε πηγή κέρδους και εσόδων. Ως προς το θέμα των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας λείπουν πολλές πληροφορίες ακόμα. Ως προς τις μεγάλες εταιρείες, οι οργανισμοί αυτοί καλά τα κατάφεραν διαχρονικά. Το πρόβλημα ανέκυψε διότι οι ρυθμίσεις απαιτούν ε, ανάληψη, ε, μάλλον ναι, ανάληψη υποχρεώσεων ως προς το κεφάλαιο. Τη στιγμή που πέφτει η πιστοληπτική ικανότητα, τότε γίνεται ε, πώληση με κίνδυνο. Αυτό σημαίνει στην Ελλάδα. Άρα πέφτουν οι τιμές και είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα, για τις επιχειρήσεις να εξεύρει χρήματα. Άρα η υπερβολική χρήση πιστοληπτικής ικανότητας στη ρύθμιση είναι ένα από τα ζητήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος ως προς την αξιολόγηση περίπλοκων προϊόντων. Εδώ ακριβώς έγκυται το πρόβλημα και το να λέμε ότι οι πληροφορίες συναλλαγής είναι διαθέσιμες σε εσά ή σε μένα, αυτό δεν θα κάνει διαφορά. Για να δούμε την αθέτηση υποχρεώσεων ως προς το χρέος, θα πρέπει να έχετε διαβάσει ένα δις πολλαπλές, ένα εκατομμύριο σελίδες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Άρα το θέμα της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αυτών των προϊόντων είναι περίπλοκο και εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό είπαμε και στο Κογκρέσο και στις ΗΠΑ. Δηλαδή αντί να έχετε μία αξιολόγηση, Νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά όταν γίνει η αξιολόγηση ο καθένας μπορεί να κινηθεί όπως θέλει. Η δεύτερη καλύτερη λύση είναι οι εκδότες να πληρώνουν για δύο αξιολογήσεις και θα αποφασίσουν ποιος οργανισμός θα τους αξιολογήσει. Ο άλλος οργανισμός ορίζεται ή τυχαία ή είναι μια δημόσια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση κάθε περίπλοκο προϊόν έχει δύο αξιολογήσεις. Εκεί που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και μια ανεξάρτητη αρχή. Και θα δούμε ποιο οργανισμό θα λάβουν σοβαρά οι αγορές. Εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αυτό δεν το ξέρετε μέσα σε έξι μήνες. Εάν υπάρχει συστημική, ένα συστημικός κίνδυνος και μεροληψία, τότε αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις από ένα πιστοληπτικό οργανισμό και στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Άρα, ως προς ένα δημόσιο οργανισμό πιστοληπτικής κανότητας, αυτό θα είναι προβληματικό, ιδιαίτερα για το κυρίαρχο χρέος, γιατί κανένας δεν θα σας πιστέψει και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος οργανισμός αξιολόγησης, για να τονίσουμε άλλες πτυχές, να δούμε τους κοινωνικούς κινδύνους, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, να έχουμε άλλη αξιολόγηση άλλων παραγόντων. Αλλά αν θέλετε μία δημόσια αρχή που να αξιολογήσει το εθνικό χρέος, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορούν να το κάνουν 27 κράτη-μέλη. Δεν μπορούν να προβούν στη σύσταση ενός τέτοιου δημόσιου φορέα. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει ή η Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν... Κοιτάξτε, δεν είχαμε σκεφτεί μια δημόσια ε, ε υπηρεσία αξιολόγησης ε, που θα ε, υπόκειται σε επιδράσεις από 27 χώρες. Σκεφτήκαμε κάτι πιο γενικό, ένα είδος ε, Ιδρύματος και ακριβώς όπως είπατε και εσείς, ένα από τα τρία και το δεύτερο θα είναι αυτό το, το ίδρυμα. Το ένα θα ήταν το Διεθνές μας Ταμείο Ναι, είναι σωστό αυτό. Η ερώτηση κυρίως βεβαίως εκτός. Το κατά πόσο το G20 και η Βασιλεία θα πρέπει να είναι δεσμευτικά βήματα. Τι πιστεύετε από αυτό Λοιπόν, νομίζω λίγο το πρόβλημα ότι εγώ ήμουν στο Βερολίνο στην ε, G20. Η G20 η ιδέα ήταν ότι δεν ήταν πολύ σημαντικό, μετά ξαφνικά έγινε σημαντικό. Τώρα με, το τρέχον, με τη τρέχουσα συνάντηση στις ε, G20 και την επόμενη θα υπάρχουν διαφορές, αποκλήσεις. Λοιπόν, ίσω θα ήταν ενδιαφέρουσα η ιδέα που προτείνεται, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω γιατί οι G20, οι βιομηχανικές χώρες και οι αναπτυσσόμενες χώρε δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χωρών που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει την Κίνα δεν είναι ενδιαφέρει μια μικρή χώρα στο νότο της Αχέλ. Και η η Βασιλεία είναι ακόμα λιγότερο αντιπροσωπευτική από ότι η ομάδα του G20. Υπάρχει βέβαια μία ε, αν θέλετε. Δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας μπορείτε να έχετε σημαντικές ε, δηλώσεις οικονομικές εφόσον δεν είναι δεσμευτικές. Εάν είναι δεσμευτικές, αυτό που θα βγαίνει από το G20 και τη Βασιλεία θα είναι αποδυναμωμένο. Ε, είναι δύσκολο να το αποφασίσει κανένας. Ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο γιατί αντιλήφθηκα ότι δεν είχα λάβει υπόψη ε, στην απάντησή μου ένα θέμα το οποίο θίξατε εσείς στην προηγούμενη ε, παρέμβασή σας. Φορολόγηση των οικονομικών συναλλαγών. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το φορολογικό φόρτο, το tax burden. Εγώ είμαι αντίθετος στη φορολόγηση των συναλλαγών, διότι αν είναι και αρκετά σημαντική, οι επενδυτές θα απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο τομέα. Και δυστυχώς αυτό είναι σημαντικό, διότι ο τομέας πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ε, προκειμένου οι τράπεζες, οι οικονομικοί, οι επενδυτικοί φορείς να αρχίσουν ε, να δραστηριοποιούνται και πάλι στον τομέα. Δεν θα πρέπει λοιπόν μόνο να έχει σημασία ως προς το tax burden, αλλά και ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει. Ορισμένες φορές υπάρχει φόρος παρακράτησης. Αλλά για τις μικροσυναλλαγές, ακόμα και κάποιος φόρος παρακράτησης ε, είναι αποθαρρυντικό στοιχείο, διότι κάποιο δεν εντάσσεται στην αγορά μετά. Ο φόρο παρακράτηση θα πρέπει να υπάρχει, αλλά για τι μεγάλε συναλλαγέ. Πακέτα ελέγχου μια επιχείρηση ή πολύ σημαντικά ή ομόλογα ε, τα οποία να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Κάτω από αυτό το όριο, όπως λέμε, the minimis not curat pretot. Από αυτά τα όρια εξελαχίστων δημιουργούνται τα σημαντικά έσοδα. Εσείς ε, ζητήσατε τρία στοιχεία, αλλά εγώ θα τα περιορίσω σε ένα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε. Να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων, είτε στην οικονομική αγορά, είτε εντός των επιχειρήσεων. Και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο βασικός όμως στόχος είναι αυτός ο οποίος είναι η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων γιατί είναι αυτός που έδωσε και το έναυσμα για την κρίση. Ε, ο εγωισμός, το γεγονός ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον για κοινά προβλήματα, αυτά που ήταν εκτός του εγώ μας ή της προσωπικότητάς μας. Αυτά που αφορούσαν δηλαδή αποκλειστικά και μόνο την επιχείρησή μας. Δεν ξέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλό θα ήταν να υπάρχει μια οδηγία ή ένας κανονισμός, δεν ξέρω, Ευρωπαϊκή Αποτροπή αποφασίσει Αυτό θα πρέπει να κάνουν ε, οι εθνικές αρχές για να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφορών. Με αυτό λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους ε, τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ που κάνατε τον κόπο να ετοιμάσετε αυτά τα έγγραφα και για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να επιστρέψετε στις χώρες σας με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ.